Λοιπόν, πρώτα-πρώτα ψηφίζουμε. Πρώτη ψηφοφορία, 14η συνεδρία των μερών της Σύμβασης για την ε, Βιοπικιλότητα. Προφορική ερώτηση προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Για το ίδιο θέμα, προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Ψηφίζουμε. And it's closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το Γενικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, όλα τα τμήματα. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 κατά, αποχές, επαλήθευση της 18, άρχεται η ψηφοφορία. And it's ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα θα ε, ψηφίσουμε για τις, ε, την διαδικασία προϋπολογισμού, για τις τροπολογίες. Θα διαβάσω μόνο τους δύο τελευταίους αριθμούς. 69 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πέρας εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Αγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και φτάσαμε στο τέλος. Ακόμα ένα θέμα μας μένει. είναι σχετικά με την απόσυρση ε, της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια ε, σχετικά με τροπολογίες 4 υπέρ κατά απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά ας Πέρας. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το υπέρ. Από 2 υπέρ. Ε, απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ηλεκτρονικά η τελική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τελειώσαμε με τις ε, ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παρακαλώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Διαφάνεια και βιωσιμότητα της εκτίμησης επικινδυνότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τροφική αλυσίδα. Εξετάζουμε το σχέδιο έκθεσης. Η κυρία Ζόμε είναι η συγγήτρια και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περιμέναμε πάνω από πέντε χρόνια μέχρι ότου τελικά μας πει η Επιτροπή εάν θα κάνει μια αναθεώρηση του, κανονισμού, του βασικού κανονισμού για την νομοθεσία των τροφίμων και αν το θεωρεί απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρούσε ότι είναι απαραίτητη ε, κάποια τέτοια αναμόρφωση του κανονισμού. Το Νοέμβριο ε, του 2017 έγινε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από διάφορες πολιτικές ομάδες και από μη κυβερνητικέ οργανώσει και εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών και τελικά καταλήξαμε σε μία ε, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών για την απαγόρευση της γλυφοσάτης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έδωσε το κίνητρο στην Επιτροπή να αλλάξει την αρχική της θέση. Με βάση την πρωτοβουλία των πολιτών, θεωρεί η Επιτροπή ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού ε, στην, ε, στα προϊόντα τροφίμων και ε, στην ομοθεσία για την τροφική αλυσίδα, ακριβώς μετά την πρωτοβουλία πολιτών για την γλυφοσάτη ε, εξετάστηκαν διάφορα θέματα όπως ε, τα θέματα διαφάνειας, τα θέματα αξιολόγησης κινδύνων, διαφάνειας κλπ. Η Επιτροπή μετά την διαβούλευση ε, είχε σχεδόν καταλήξει το αποτέλεσμα και φάνηκε σαν να ήταν έτοιμη η άποψη της Επιτροπής ακόμη και πριν την διαβούλευση η οποία ήταν πολύ σύντομη. Όπως είπαμε, η Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Γλυφοσάτη έκανε την Επιτροπή ε, να ε, αλλάξει θέση και από το 1 εκατομμύριο υπογραφών οι 600.000 προέρχονται από ένα και μόνο κράτο μέλο. και αυτό μου φαίνεται κάπως περίεργο. Αυτό δείχνει και πόσο ε, αντιπροσωπευτική ήταν αυτή η Πρωτοβουλία Πολιτών ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απλώς μια παράπλευρη παρατήρηση. Μου φαίνεται ε, ότι ε, δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε πώς η Επιτροπή αποφασίζει να περάσει σε νέους κανόνες με βάση μόνο αυτά τα στοιχεία. Κατά την αξιολόγηση καταλληλότητας του βασικού κανονισμού, την REFIT, ε, ε, η ισχύουσα νομοθεσία, ο βασικός κανονισμός, είχε θεωρηθεί ότι είναι ε, κατάλληλος. και με τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Προστασία των Τροφίμων πάλι τα, αποτελέσματα ήταν ε, ε, ικανοποιητικά και η Επιτροπή είχε καταλήξει ε, μετά την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων ότι η refit του βασικού κανονισμού, η αξιολόγηση καταλληλότητας ήταν επαρκής μετά την πρωτοβουλία πολιτών ε, για την ε, γλυφοσάτη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εξέτασε όλες τις εναλλακτικές λύσεις και υπάρχει μια επιτροπή η οποία συστάθηκε και βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία. Είναι η διαδικασία της δημοκρατικής διαμόρφωσης άποψης, την οποία όμως τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να αγνοεί και δεν περιμένει την ολοκλήρωσή της και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Επιπλέον, βρισκόμαστε λίγο πριν τις, Ευρω... τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καν τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τη δέουσα επιμέλεια, με την πρόταση της Επιτροπής και να ζητήσει και τη γνώμη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων μας θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πολύ μικρό χρονικό περιθώριο που δεν μας αφήνει καθόλου τη δυνατότητα να καλέσουμε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες τώρα και ε, μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές. Και το Συμβούλιο Υπουργών εξεπλάγει, όπως και εμείς, λόγω της ταχύτητας με την οποία η Επιτροπή θέλησε να διεκπαιρεώσει αυτή τη διαδικασία. Μέχρι τον Νοέμβριο αναμένεται η κοινή θέση του Συμβουλίου και μένουν μόνο πέντε εβδομάδες ε, για τον τριμερή διάλογο μέχρι, τα, ε, μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων ε, και τέλη Ιανουαρίου πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τον τριμερή διάλογο. Το αργότερο τον Μάρτιο συγγνώμη, του 2019 πρέπει να έχουμε ψηφίσει το θέμα στην Ολομέλεια γιατί έχουμε να ασχοληθούμε και με τα θέματα του Brexit και με... να ακολουθούν και οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπουμε ότι η Επιτροπή σε αυτή την περίπτωση προσπαθεί να ε, βιάσει πολύ τα πράγματα και είναι εντυπωσιακή αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής, την οποία σημειώνει και το Συμβούλιο. Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι αυτό το θέμα ε, φτάνει τώρα, λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, και αυτό επηρεάζει οπωσδήποτε και ε, τις εργασίες που γίνονται και το αποτέλεσμα ε, των ε, εργασιών μας. Δεν υπάρχει αξιολόγηση των επιπτώσεων σε αυτή την έκθεση της Επιτροπής. Αυτό είναι αδιανόητο. Θα έπρεπε να εξεταστούν οι διάφορες επιλογές και για το χρονικό σημείο στο οποίο φτάνει μια τέτοια πρωτοβουλία της Επιτροπής γιατί η χρονική στιγμή μπορεί να έχει δραματικές επιπτώσεις ε, στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιριών. Θα πρέπει να εξεταστούν διάφορα οικονομικά μοντέλα να έχουν κάποιο ρόλο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων. Δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία και θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη της. Υπάρχουν νέοι κανόνες για τη διαφάνεια, για τους οποίους έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις η ΕΦΣΑ, η Ευρωπαϊκή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ήδη δημοσιεύει στοιχεία ε, και ισχύει ο κανονισμός ε, για την πρόσβαση σε έγγραφα. Θα πρέπει να ισχύσουν οι ίδιες διατάξεις όπως ε, ισχύουν για τη διαφάνεια στους άλλους εξωτερικούς οργανισμούς, αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ζητείται η κοινοποίηση πληροφοριών τη στιγμή που υποβάλλονται οι φάκελοι αίτησης ε, ε, έγκρισης ε, πριν ολοκληρωθούν οι τεκμηριωτικές μελέτες. Αυτό ανοίγει το δρόμο σε μια πειρατεία ιδεών. Κάποιοι ανταγωνιστές ε, στην Κίνα, παραδείγματο χάρη, θα μπορούσαν μέσω του διαδικτύου να ενημερωθούν για το τι αιτήσει έγκριση έχουν υποβληθεί και να αντιγράψουν πιθανέ καινοτομίε ευρωπαϊκών εταιριών, ε, οι οποίε έχουν υποβάλει αίτηση αλλά δεν έχουν ακόμη πάρει την άδεια εφόσον ε, συνεχίζονται, συνεχίζεται η διεξαγωγή των ε, εκθέσεων τεκμηρίωσης διαδικασία ε, έγκρισης των αιτήσεων από την ΕΦΣΑ διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα και όσο διεξάγονται αυτές οι εργασίες ε, από την ΕΦΣΑ μπορούν οι ανταγωνιστές να αντιγράψουν το προϊόν ε, πριν ο Ευρωπαίος κατασκευαστής αποκτήσει άδεια για το προϊόν. Αυτό αποτελεί ε, σπατάλη χρόνου και πόρων, ε, εκτός από το ότι πλήττει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν γίνεται η δημοσίευση ε, θα πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει η επιστημονική άποψη της ΕΦΣΑ, όταν ε, η ΕΦΣΑ είναι έτοιμη να δημοσιεύσει ε, το αποτέλεσμά της βάσει των μελετών τεκμηρίωσης. Αυτό ακολουθείται και από, τις ε, άλλες, από τους άλλους αποκεντρωμένους οργανισμούς, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Ουσιών και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Επίσης, ε, δεν καταλαβαίνω γιατί να ισχύουν πιο ε, αυστηρές διατάξεις για την αξιολόγηση των κινδύνων, γιατί υπάρχει και η φάση αξιολόγησης, υπάρχουν οι φάσεις της αξιολόγησης κινδύνων, της διαχείρισης κινδύνων και της ε, ανακοίνωσης και ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους. Γιατί να είναι λοιπόν μόνο η φάση της εξέτασης των κινδύνων αυτή στην οποία θα ισχύουν οι πιο αυστηρές διαδικασίες θα μπορούσαν να επηρεάζονται πολλές αποφάσεις από πολιτικές ε, προσπάθειες των κρατών μελών αν ε, στην ΕΣΑ έχουν μεγάλη επιρροή τα κράτη-μέλη. Προτείνεται επίσης ε, μιας και στην ΕΦΣΑ εξετάζονται πολλού είδους, προϊόντα και τρόφιμα και πρόσθετα ε, και ε, ε, μέσα φυτοπροστασίας δεν εκπροσωπούν δεν μπορεί να εκπροσωπούνται ε, μόνο με μονομένη κλάδη. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μόνο ένας ε, εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ε, ΕΦΣΑ, αλλά τουλάχιστον δύο, γιατί θα πρέπει να εκπροσωπείται αφενός μεν ο τομέας τροφίμων και προσθέτων, αφετέρου δε ο τομέας των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και μέσων φυτοπροστασίας η Επιτροπή νομίζω ότι έχει υπερβεί ε, το απαιτούμενο τον απαιτούμενο βαθμό εγγύσεων που απαιτούνται όταν ζητά εκπροσώπους ε, από κάθε κράτος μέλος ε, και για τους εμπειρογνώμενους που απαιτεί η ΕΦΣΑ αν ε, ε, όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν δική τους πρόσκληση ενδιαφέροντος για να επιλέξουν εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα σταλούν στην ΕΦΣΑ, αυτό δεν θα είναι προς συμφέρον της ΕΦΣΑ, διότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια ανταλλαγή ε, εκπροσώπων των κρατών μελών και εμπειρογνωμόνων ανάλογα και με τα θέματα τα οποία εξετάζονται. Δεν εξοικονομούμε πόρους, αλλά αντιθέτως δημιουργούμε μεγαλύτερη ε, γραφειοκρατία αν θα πρέπει να εναλλάσσονται οι εκπρόσωποι των κρατών μελών για τα διάφορα θέματα που εξετάζει η ΕΦΣΑ. Θα μπορούσα ε, ως ε, συμπέρασμα να σας πω τα εξής. Έχω κάνει κάποιες τροπολογίες και μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου που είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ε, θα προετοιμάσω και άλλες τροπολογίες. Δεν είχαμε μεγάλο χρονικό διάστημα ούτως ή άλλως. Και είμαι βέβαιη ότι και οι συνάδελφοι θα έχουν πολλές τροπολογίες. Έχουμε ήδη μια πρόγευση αυτών ε, τα οποία ε, θα ακολουθήσουν. Δεν θα συμφωνήσουμε μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων, αλλά αυτό είναι και αναμενόμενο στην Επιτροπή Γιούρι και Αγκρή έχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες ε, πολύ συχνά ταυτίζονται, ε, αλλά πολλές φορές ε, δεν υπάρχουν και πλήρης επεξηγήσεις των τροπολογιών για να, να καταλάβω και εγώ την πρόθεση πίσω από την τροπολογία. Θα το συζητήσουμε όμως με τους εισηγητές. Πάντως και οι δύο επιτροπές θεωρούν την σύμβαση του Όρχους ως απαραίτητη βάση για τα όσα θα συζητήσουμε. Και εδώ έχω και άμεσα ένα ερώτημα προς την Επιτροπή, διότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς αξιολογεί από νομικής πλευράς αυτές τις απαιτήσεις η Επιτροπή και τι θα κάνουμε με τον τομέα των ε, ε, τροφίμων, γιατί αυτά είναι για τον τομέα των ε, φυτοφαρμάκων, θα πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε και για τον τομέα των τροφίμων. Παρακαλώ τους συναδέλφους στις τροπολογίες τους να εστιαστούν μόνο στα σημαντικά σημεία. Να εστιαστούμε στην πρόταση της Επιτροπής και να μην επεκταθούμε σε άλλες ε, τροπολογίες για διαφορετικά προϊόντα. Λόγω της χρονικής πίεσης δεν θα γίνουν αποδεκτές τροπολογίες που αφορούν άλλους τομείς πέραν αυτών που ε, τίθενται από την Επιτροπή στην πρότασή της. αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλει και άλλες τροπολογίες πέραν του πεδίου που καλύπτεται από την πρόταση της Επιτροπής, θα ε, αποτύχει η προσπάθειά μας στο Συμβούλιο, θα απορριφθεί από το Συμβούλιο. Μιλάμε για τους κανόνες διαφάνειας, αλλά δεν θέλουμε να επεκταθούμε σε όλους τους τομείς. Ξέρω ότι είναι μεγάλη πρόκληση να πούμε αυτό το οποίο θέλουμε και για τους άλλους τομείς, αλλά δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Σας παρακαλώ λοιπόν δείξτε αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τις τροπολογίες. Θα πρέπει λόγω της πίεσης χρόνου να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους πολίτες της Ευρώπης και δεν θέλουμε να δώσουμε λάθος μήνυμα πριν από τις εκλογές. Αν αποτύχουμε με αυτό το θέμα στην επόμενη θυμία, στην επόμενη θητεία, συγγνώμη, θα προκύψει κάποια καινούργια πρόταση της Επιτροπής προς την ίδια κατεύθυνση. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τώρα με την πρόταση αυτή να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο οφείλουμε στους πολίτες της Ευρώπης, μεγαλύτερη διαφάνεια, μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τους κοιόδης ηγητές τώρα, οι οποίοι θα το λόγο. Σας παρακαλώ λίγο, έχετε κατά νου το χρόνο, μην ε, υπερβείτε τα όρια, διότι έχω και ένα μακρύ κατάλογο μιλητών που θέλουν το λόγο. Ο κύριος Πότς καταρχάς. Ε, ευχαριστώ. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε και μπορεί να σας εκπλήξει μεν, αλλά στην ουσία συμφωνώ μαζί της σχεδόν σε όλα. Οι πιο ε, βαριές επικρίσεις είναι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν θα είμαι λίγο πιο σκληρός από την εισηγήτρια. Τις δημόσιες διαβουλεύσεις τις έχει κάνει ε, ουσιαστικά κομμωδία και εμεί είμαστε απλώς παλιάτσι διότι έχουμε ελάχιστο χρόνο να διορθώσουμε όλα τα λάθη τα οποία ε, περιλαμβάνονται στην πρόταση. Ε, μου θυμίζει λίγο μια κατάσταση σαν αυτή που είχαμε το 2014 ε, όταν ε, συζητούσαμε τα αλόχθονα επιθετικά είδη. Ε, χαίρομαι που η συγγήτρια έκανε κάποιες προτάσεις τροπολογίας, ε, κυρίως εναντίον όσων θέλουν να ε, προσβάλλουν τις μελέτες όσον αφορά τον διορισμό στα επιστημονικά πάνελ, ε, τα θέματα της εμπειρογνωμοσύνης. Συμφωνώ μαζί της όσον αφορά την περισσότερη διαφάνεια στις αποφάσεις και όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου, σίγουρα ε, τη δημοσίευση των, πρακτικών ε, και των ψηφοφοριών, των συνεδριάσεων, όλα αυτά είναι ε, πράγματα με τα οποία συμφωνώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υποσχέθηκε ότι στην πρότασή της θα εγγυηθεί μεγαλύτερη διαφάνεια για τον κίνδυνο στην διατροφική αλυσίδα. Ε, έχω κάποιες αμφιβολίες, διότι η πορεία που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πιστεύω ότι είναι προς όφελος της όλης διαδικασίας. Για παράδειγμα, εγώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς ε, για ποιο λόγο αντικαθίσταται ο κατάλογος ε, πληροφοριών που έχουμε αυτή τη στιγμή με το λεγόμενο κατάλογο πληροφοριών που μπορεί να είναι και εμπιστευτικέ, εκτός και αν υπάρχει κάποιο ε, ε, ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον. Φαντάζομαι τέτοια συζήτηση. Τι σημαίνει ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον. Υπάρχει ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση. Ε, και αυτές οι πιθανόν ε, ε, εμπιστευτικέ πληροφορίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο ή όχι. Σε αυτές λοιπόν τις πιθανόν εμπιστευτικέ πληροφορίες κατά πάσα πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για την αξιολόγηση του κινδύνου και για το περιβάλλον και για τη δημόσια υγεία. Παραδείγματο χάρη οι πληροφορίες όσον αφορά τη σύνθεση των φυτογειονομικών προϊόντων. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, μια νομοθεσία η οποία θα έπρεπε να εγγυάται περισσότερη διαφάνεια εδώ να κάνει ένα βήμα προς τα πίσω. Πολλές από αυτές τις πληροφορίες λοιπόν στον κατάλογο ε, θα διαγραφούν κατά πάσα πιθανότητα. Η συγγήτρια είπε ότι πρέπει να σεβαστούμε ε, την οδό που με υπερεπτικό τρόπο μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν θα υπάρχει χρόνος για να ε, μπορέσουμε να έχουμε αξιολόγηση επιπτήσεων. Αν υποχρεωθούμε όμως να σεβαστούμε όλα αυτά, τότε θα πρέπει να προετοιμάσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ένα κατάλογο οριζόντιων πληροφοριών. Πληροφορίες οι οποίες ε, εάν δεν δημοσιοποιηθούν, θα είναι εις βάρος ε, του δημοσίου συμφέροντος. Ελοχεύει όμω ο κίνδυνο η διαφάνεια να είναι μικρότερη από αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε η συγγήτρια, ε, είναι να μην ε, ε, είναι εις βάρος ε, της πρόσβασης των ε, πολιτών σε πληροφορίες στο νέο καθεστώς. Διότι ορισμένες φορές είναι η μόνη διέξοδος που έχουμε. Από την άλλη βέβαια δεν θα πρέπει να εμποδίζουμε και τον κλάδο να καινοτομεί ε, και φυσικά να ε, βοηθήσουμε και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν. Επίσης να πω είμαστε δυσαρεστημένοι και με την αιτιολογική σκέψη 27, διότι τα θέματα της διαφάνειας όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τον 178 του 2002. Εδώ η πρόταση λοιπόν θα πρέπει σίγουρα να τύχει επανεπεξεργασία για να μην ε, προσβάλλουμε το δικαίωμα των πολιτών που απορρέει από τον κανονισμό του 2001 για την ε, πρόσβαση ε, σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων και επίσης να μην τεθεί και ένα αμφιβόλο η σύμβαση του άρχους. στην ουσία η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε πάρα πολύ βεβαιασμένα. Επίσης, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κλάδου. Ε, δεν ξέρω, ίσως θα ήταν καλύτερη η λύση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος προστατεύει τα λεγόμενα raw data, τα ε, ανεπεξέργαστα στοιχεία δηλαδή, ε, από όσους θέλουν να κάνουν εμπορική χρήση αυτών των στοιχείων. Ίσως αυτή θα ήταν μια καλύτερη προσόγγιση, διότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Τώρα, μελέτες επαλήθευσης, ε, σίγουρα είναι μια θετική πρόταση αυτή. Θα μπορούσαν ίσως να λύσουν και το πρόβλημα της ανεπάρκειας κάποιων στοιχείων, αλλά οι μελέτες αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί της αρχής της προφύλαξης. Και επίσης δεν θα πρέπει να τις εκμεταλλεύεται ο κλάδος ε, για να ε, κερδίσει χρόνο για να επιλύσει ε, κάποια προβλήματα τα οποία θεωρούνται προϊόντα υψηλού κινδύνου. Και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή τα κενά τα οποία επεσήμανε ο ΕΦΣΑ στις γνωμοδοτήσεις του, βάσει των οποίων υπάρχουν ουσίες στην αγορά παρά το γεγονός ότι λείπουν στοιχεία για τον καθορισμό της ποιότητας αυτών των ουσιών. Ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται να μιλάτε τόσο πολύ για το θέμα αυτό. Σας παρακαλώ, ακόμα και αν είστε σκιώδης συζητητής, μην υπερβείτε τα πέντε λεπτά. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γκέρκε. Ja, herzlichen Dank. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την ε, πλήρεστατη έκθεση. Εδώ δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ε, πολιτική καταναλωτών. Θέλουμε να έχουμε στοιχεία τα οποία θα είναι ελέγξιμα. Και χρειάζεται ε, έλεγχος της διαφάνειας, τον οποίο ε, να μην επηρεάζουν ε, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες σε βαθμό που να μην υπάρχει διαφάνεια για τους ε, καταναλωτές. Όσον αφορά την ΕΦΣΑ, πάρα πολλά στοιχεία ετέθησαν προς, προς εξέταση και εξετάστηκαν πάρα πολλά στοιχεία, αλλά όπως είπατε ήταν πολύ περιορισμένο το χρονικό διάστημα. για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη εξέτασης όλων των ε, στοιχείων. Μιλάμε για τρόφιμα, μιλάμε για προστασία και επομένως ε, συμφωνώ με την κυρία Ζώμε ότι θέλουμε να έχουμε ε, καλύτερη πρόταση από την Επιτροπή, να μένουμε μια καλύτερη πολιτική από την Επιτροπή και όσον αφορά τις ε, πολυεθνικές εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χόσλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε μία πρόταση της Επιτροπής που αρχικά την είδαμε με χαρά. Θεωρήσαμε ότι θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια, θετικό αυτό. Μετά την ιστορία με τη γλυφοσάτη κάτι έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουμε. Και μετά την πρωτοβουλία των πολιτών για τη γλυφοσάτη ε, είπαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν τα πράγματα όσοι είχαν στο παρελθόν. Όταν μπήκαμε όμως στις λεπτομέρειες της πρότασης της Επιτροπής απογοητευθήκαμε. υπάρχουν ε, σημεία τα οποία μας δημιούργησαν ε, έλλειψη εμπιστοσύνης και αναρωτηθήκαμε αν η πρόταση της Επιτροπής είναι όντως ε, μια προσπάθεια βελτίωσης ή αν είναι ένα βήμα προς τα πίσω. Και είπαμε όλοι ότι είναι λυπηρό ότι μας έθεσε η Επιτροπή σε τόσο μεγάλη πίεση χρόνου. Γιατί θα έπρεπε τόσο γρήγορα να ανταποκριθούμε ε, στην ε, πίεση αυτή της Επιτροπής. Θα πρέπει πριν από το τέλος της θητείας μας να το ολοκληρώσουμε ε, αλλά τουλάχιστον να πρόκειται για κάτι που θα βελτιώσει τη διαφάνεια και εξετάζοντας την πρόταση της Επιτροπής έχουμε αρκετές παρατηρήσεις. Η δημιουργία ενός δημοσίου μητρώου είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε και η δημοσίευση των στοιχείων επίσης είναι θετικό. Η δημοσίευση των ανεπεξέργαστων δεδομένων καταρχήν είναι καλές προτάσεις. Δημοσίευση όταν υποβάλλεται η αίτηση στην ΕΦΣΑ. Αλλά... Ε, βλέπουμε με την εξέταση της πρότασης της Επιτροπής ότι δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια όπως ισχυρίζεται η Επιτροπή. Υπάρχουν αντιφάσεις και με τη σύμβαση του Όρχους και μας δημιουργεί ε, πραγματικά δυσπιστία. Χρειάζεται τροποποίηση η πρόταση της Επιτροπής σε συγκεκριμένα σημεία. θα πρέπει να δημιουργείται ένας ε, κατάλογος πληροφοριών οι οποίες πρέπει να παραμένουν ε, απόρριτες ε, και όταν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα πρέπει να, είναι, να εξετάζεται το κατά πόσο είναι δυνατόν να δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες. Το άρθρο 39 ε, για την πρόσβαση σε δεδομένα ε, θα πρέπει να ε, συμβαδίζει με τη σύμβαση του Όρχους. Δεν θέλουμε να περιορίζεται το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση σε δεδομένα, αλλά θέλουμε να βελτιωθεί η σχετική διάταξη. Ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Ζόμε, στο οποίο έχουμε κάπως διαφορετική άποψη. Θέλουμε συμμετοχή των κρατών μελών στις, ε, ε, στη διαδικασία εξέτασης της ΕΦΣΑ, αλλά δεν συμφωνούμε με την ε, εκπροσώπηση του κλάδου. Θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το θέμα αυτό και να δούμε κατά πόσο θέλουμε εκπρόσωποι των εταιριών να συμμετέχουν. Και όσον αφορά τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, ε, το ανέφερε και η κυρία Ζόμεχ, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να γίνεται ένας ανοιχτός διαγωνισμός και ανοιχτός διορισμός των επιλεγόντων. των επιλεχθέντων, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν όλες οι πολιτικές ομάδες θα συμφωνήσουν για αυτά τα θέματα, αλλά και από τη συζήτηση στην Επιτροπή Γεωργίας πρέπει να δούμε ε, αν έχουμε την κοινή γραμμή, γιατί έχουμε μια ερώτηση προς την Επιτροπή ε, ε, και μπορεί η Επιτροπή να άρει την έλλειψη σαφήνειας που υπάρχει. Ελπίζουμε ότι θα συνεργαστεί η Επιτροπή, διότι αυτό το οποίο ε, είναι ενδιαφέρον και για την κοινή γνώμη είναι αν αυτή η πρόταση της Επιτροπής όντως μας οδηγεί ε, σε μια καλύτερη κατάσταση ε, ή αν είναι ένα βήμα προς τα πίσω. Αν δίνουμε, ένα, αν δίνουμε μεγαλύτερες εξουσίες στη βιομηχανία αντί να προστατεύουμε περισσότερο τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάζελκαμπ. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση, η πρόταση της Κομισιό θέλει να κάνει την διαδικασία πιο διαφανή. Είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν είναι εύκολο βεβαίω εκ πρώτη όψεω. Όταν κοιτάξει κανείς λεπτομερώς το περιεχόμενο της έκθεσης, βλέπετε ότι αν διατηρηθεί το κείμενο ως έχει, οι προτινόμενοι νέοι κανόνες θα οδηγήσουν ίσως σε λιγότερη διαφάνεια από ό,τι έχουμε σήμερα. και θα δώσω μερικά παραδείγματα. Οι περισσότερες πράξεις που θα αντικατασταθούν περιλαμβάνουν καταλόγους πληροφοριών που θεωρούνται περίπου εμπιστευτικές και οι κατάλογοι αυτοί θα αντικατασταθούν με καταλόγους που θα θεωρηθούν ε, εμπιστευτικοί ε, εάν ε, θεωρηθεί κατάλληλο. Και έχω μια ερώτηση στην Κομισιόν. Στόχος είναι να μελιορέσετε την διαφάνεια γιατί Πιστεύετε ότι οι φυστάμενοι κατάλογοι δεν θεωρούνται εμπιστευτικοί. Θεωρείτε ότι αν κρατήσουμε αυτούς τους καταλόγους ε, θα, θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια. Υπάρχουν νέες διατάξεις ότι η αποκάλυψη επιστημονικών ε, στοιχείων και μελετών με άδεια δεν ε, θα θίξει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τα οποία υπάρχουν, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το άρθρο 38 θέτει μια νέα βάση ε, για να ε, απορρίψει την πρόσβαση σε ε, πληροφορίες λόγω δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Δεν θα μιλήσω πολύ για την σύμβαση Άρους, αλλά έχω μια ερώτηση στην Κομισιόν. Θέλετε περισσότερη διαφάνεια γιατί περιλαμβάνεται ε, το 36α ε, θέτοντας ένα αμφιβόλο την πρόσβαση ε, σε κείμενα, διότι η πρόταση είναι, αν θέλετε, προδραστική αποκάλυψη πληροφοριών και μελετών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να περιορίζεται το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα. Ένα τελευταίο σημείο σχετικά με το σχέδιο της κυρίας Σόμερ που περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία, αλλά το κρίσιμο σημείο για μένα είναι ότι όλο το σχέδιο έκθεσης έχει ε, βασική αντίρρηση στην ε, δημοσίευση ε, των στοιχείων παρά μόνο όταν η αρχή έχει εκφέρει τη γνώμη της. Και αυτό είναι αντίθετο προς όλες τις προσπάθειες διαφάνειας, διότι οι ανεξάρτητοι θα μπορούν να ελέγξουν μόνο όταν θα έχουν τα στοιχεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ευκαιρία για ανεξάρτητη εξέταση επιστημονική προ, ε, προτού. Και αυτές είναι οι αντιρρήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εμείς ε, είμαστε υπέρ και είμαστε ικανοποιημένοι που υπάρχει αυτή η πρόταση. Ακούστηκε ε, πολύ το θέμα της ε, ανανέωσης της άδειας της γλυφοσάτης και της ανανέωσης των αδειών προϊόντων γενετικώς τροποποιημένων. Επομένως, ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα ότι ε, θα πρέπει να, διότι θα γίνεται μια πρόταση μεταρρύθμισης του τρόπου εξέτασης αυτών των προϊόντων. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο έχουν ε, ζητήσει οι πολίτες και το αίτημα της διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε εδώ πέρα να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των κινδύνων για να μην έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ε, πρέπει να το αλλάξουμε σε μερικά χρόνια. Και αναρωτιέμαι και πόσες από αυτές τις μελέτες ε, οι οποίες θα ζητηθούν ε, θα δημοσιοποιούνται από εκεί και πέρα. Αυτή τη στιγμή ο κλάδος δεν έχει κανένα όριο. Μπορεί να υποβάλει αιτήματα εμπιστευτικότητας χωρίς περιορισμό. Ε, και επίσης ε, τι θα πρέπει να κάνουμε για να γνωρίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία. Εάν, όπως έλεγε η κυρία Χάζενκαμπ, ο στόχο είναι να αυξήσουμε τη διαφάνεια, όλοι αυτοί οι περιορισμοί στην πραγματικότητα απλώ περιορίζουν τη διαφάνεια. Όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΦΣΑ, μεταξύ των καθηκόντων του υπάρχει σαφέστατα και είναι γραμμένο ο ε, διορισμός των μελών και του Προέδρου της επιστημονική Επιτροπή και των Εμπειρογνωμόνων. Πώς μπορεί λοιπόν ε, να μην έχει αντίκτυπο ε, στην ανεξαρτησία του επιστημονικού έργου ε, αυτή η δυνατότητα. Επίσης, η νέα πρόταση ε, προτείνει αύξηση των μελών και θα υπάρχουν εκπρόσωποι από κάθε κράτο μέλο πέραν των εκπροσώπων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ συμφωνώ με τον συνάδελφο από του Πρασίνου ότι απαιτείται τουλάχιστον παρουσία δύο εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι θέση έχουν τα κράτη-μέλη ε, και κλεισμένων των θυρών και πώ ψηφίσουν για ουσιαστικά ζητήματα ε, για τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Τέλος, κάτι για τον προϋπολογισμό της ΕΦΣΑ. Είναι σαφές ότι αν όλοι αναγνωρίσουμε την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας και της βελτίωσης της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου, πρέπει να προσαρμοστεί και ο προπολογισμό ε, της ΕΦΣΑ, γιατί αλλιώ ε, τα πάντα θα παραμείνουν ένα ουτοπικό όνειρο. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές και ξεκινάμε με την κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω πολύ χρόνο, θα είμαι σύντομη. Καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Σόμερ και να πω ότι συμφωνώ σε πολλά. Πραγματικά υπάρχει ταύτιση απόψεων. Και κάποια γενικά σχόλια. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αφήσει ε, το, η κληρονομιά της ε, με αυτή την πρόταση, αλλά αν είχαμε μια πιο φιλόδοξη πρόταση, ε, θα είχαμε τον, ε, τη μεταρρύθμιση του 178 του 2002. Δεν πρέπει να αναλύσουμε μόνο τα θέματα της ΕΦΣΑ, αλλά και τα δίκτυα εκτάκτου ανάγκης, το θέμα της ε, διατροφής ε, είναι ε, πράγματα τα οποία βρίσκονται επιτάπητο. Θα έπρεπε όμως να γίνει με μεταρρύθμιση. Δεν ξέρω, δεν είναι μεταρρύθμιση αυτό, είναι αναθεώρηση στην πραγματικότητα. Το σχέδιο πρότασης ε, φαίνεται ότι έχει μια επίγουσα πολιτική ανάγκη και αυτό είναι σαφές και αυτό δεν είναι καλό. Αυτά που αναφέρονται στις αιτιολογικές και εκθέσεις ε, για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών για τη γλυφοσάτη το αποδεικνύουν. Στην ουσία είναι ένας κανονισμός ο οποίος δεν αναθεωρεί, δεν μεταρρυθμίζει, απλώς αναθεωρεί εννέα νομικά κείμενα και αυτό δεν είναι θετικό. Συμφωνούμε με τους βασικούς στόχους, να διευκρίνουμε τους κανόνες διαφάνειας, να έχουμε αντικειμονικότητα, να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση, να, μειώσουμε, να βελτιώσουμε την αριστεία κλπ. Όλα αυτά είναι ευγενεί στόχοι και τους ε, υποστηρίζουμε. Αλλά υπάρχει και το θέμα των μελετών Μονσάντο και της Γλυφωσάτης και την ανάγκη να προσελκύσουμε επιστήμονες ε, και να ανοίξουμε την εύσα σε όλα τα κράτη-μέλη, να υπάρχει καλύτερο συντονισμός ε, με τα κράτη-μέλη για να αποφύγουμε θέματα ε, ε, και προβλήματα επικοινωνία. Όσον αφορά τα άρθρα, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να υποστηρίξω την κυρία Ζόμερ και να πω ότι όσον αφορά ε, τους εκπροσώπους, καλό είναι να έχουμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τον κλάδο, τους γεωργούς κλπ. Αλλά δεν υπάρχουν εκπρόσωποι τη αλυσίδα διανομής, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, διατροφικής αλυσίδας και φυσικά βοηθούν ιδιαίτερα στην όλη διαδικασία. Οι εμπειρογνώμονες, ε, ε, δύο από κάθε κράτος μέλος, και λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι η ΕΦΣΑ πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και να σταματήσει να προσπαθεί να είναι ένας καθαρά διοικητικός οργανισμός με πολύ αυστηρούς κανόνες. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Θα ήθελα να πω το εξή. Υπάρχουν θετικά στοιχεία μεν, αλλά εγώ πιστεύω ότι ε, δεν είναι πλήρης μεταρρύθμιση, επαναλαμβάνω, είναι απλώς μια αναθεώρηση και ίσως στο νομοθετικό σχέδιο θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στοιχεία τα οποία απουσιάζουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο συντονισμό, στον οποίο θα πρέπει η ΕΦΣΑ να είναι πολύ πιο δραστήρια και να λαμβάνει υπόψη τη τον ε, πολίτη. Να υπάρχει μια εσωτερική αρχή που θα λαμβάνει υπόψη της ε, τα θέματα της διατροφικής ασφάλειας και της υγείας και να υπάρχει και συμμετοχή και συνένεση ε, των ε, διαφόρων παραγόντων και να μην υπάρχουν και τα λεγόμενα fake news, οι ψευδείς ειδήσει και να μαθαίνει την αλήθεια ο καταναλωτής. Ξέρω ότι υπάρχει έλλειψη χρόνου και ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε το χρονοδιάγραμμα, αλλά πιστεύω ότι λόγω χρονικών περιορισμών δεν έχουμε το ε, περιθώριο να κάνουμε κακές επιλογές και πιστεύω ότι καλύτερο θα ήταν να μην έχουμε καθόλου πρόταση από το να έχουμε μια τόσο κακή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ομαζή. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θεωρούμε ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και κυρίως των φυτοφαρμάκων και της γλυφοσάτης είναι σκάνδαλα, σκάνδαλα υγειονομικά και σε αυτά προστίθενται και σκάνδαλα δημοκρατίας. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σκάνδαλα τώρα. Υπάρχει μια τάση ιστορική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιφρονεί ε, το Κοινοβούλιο. Αλλά όταν δεν μπορούμε ε, να έχουμε σεβασμό, μας περιφρονούν. Και υπάρχει μια τάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι γελίο. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου αποφασίσαμε όταν ε, είχαμε το σκάνδαλο γλυφοσάτης να έχουμε μια επιτροπή φυτοφαρμάκων, τζιζανιοκτώνων. Εγώ είμαι στην επιτροπή αυτή μέλος και εργαζόμαστε για περισσότερη διαφάνεια, για λιγότερη εμπιστευτικότητα, για τον τρόπο με τον οποίο θα είναι ε, δυνατόν να μην υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στην Κομισιόν και τα λόμπι και να γίνει μια σοβαρή εργασία για όλο αυτό το φάκελο των φυτοφαρμάκων και εδώ η Κομισιό μας ε, παρεμποδίζει με μία πρόταση που είναι κατακριτέα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή, τουλάχιστον αυτό θα πω σήμερα το απόγευμα ε, στην Επιτροπή Φυτοφαρμάκων. Θα πρέπει να διαλύσουμε τότε αυτή την Επιτροπή. Ή αλλιώς η η δικη μας η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν κάνει αυτή την πρόταση τροπολογιών σε σχέση με τα όσα προτείνει η Κομισιό. Είναι ή το ένα ή το άλλο, διότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο ε, δίνεται δίκιο ε, όλοι όσοι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιφρονεί το δικό μας κοινοβούλιο. Τούτων λεχθέντων, όταν βλέπει κανείς αυτή την πρόταση, βλέπετε ότι κάτω από ένα λούστρο περισσότερης ε, διαφάνειας έχουμε λιγότερη διαφάνεια. Κάτω από αυτή την, ε, τη βιτρίνα ε, θα έχουμε περισσότερα μυστικά, περισσότερη εμπιστευτικότητα και έτσι έχουμε πρόβλημα με την ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών θεσμών. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής. Τελευταίο πράγμα. Το λέω και το επαναλαμβάνω σήμερα. Η ιστορία θα καταδείξει ότι το θέμα της γλυφοσάτης δεν ε, και άλλων ε, φυτοφαρμάκων, αλλά κυρίως της γλυφοσάτης, θα αναγνωριστεί ως ένα από τα σοβαρότερα υγειονομικά σκάνδαλα στην ιστορία της Ευρώπης. Και εμείς συνεδριάζουμε εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε ευθύνη, έχουμε καθήκον να πούμε στους πολίτες ότι δεν είναι προστατευμένοι, ότι υπάρχουν ε, συνωμοσίες με τα λόμπι και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια αντιεξουσία, θα πρέπει να έχουμε θέσεις στεναρές, αυστηρές και το πρώτο πράγμα είναι να υπάρχει σεβασμός για την δημοκρατία, διότι ζούμε τώρα μια φάρσα δημοκρατική. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Λάβια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της και να συμφωνήσω μαζί της όσον αφορά τις ανησυχίες της για ε, πάρα πολύ στενά περιθώρια εντός των οποίων θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει το θέμα. Πιστεύω ότι η πρόταση που κάνατε είναι πολύ καλύτερη από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως θα σταθώ σε δύο πτυχές. Ε, μία πτυχή η οποία έχει σχέση με τη λεγόμενη διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών. Διότι δεν θα θέλαμε για να αυξηθεί η διαφάνεια, να μειωθεί η ανταγωνιστική δυνατότητα του συστήματός μας με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει και τις επιχειρήσεις να αποσύρουν πλήρως ένα φάκελο για να έχουν έλεγχο κάποιων πληροφοριών. Και η δεύτερη πτυχή είναι μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή ε, την οποία επισημαίνω και παρουσία και της ΕΦΣΑ και της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, διότι αυτοί οι μηχανισμοί δεν επιτρέπουν και δεν θα επιτρέψουν να βελτιώσουμε τη διαφάνεια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και το δίνω με βάση μια ουσία, την πρόσφατη περίπτωση της επιστημονικής γνωμοδότησης των παραγόγων ε, ανθρακ κινήνων που χρησιμοποιούνται σε διάφορες ουσίες όπως αποκαλούνται. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες χωρίς να έχουν υπάρξει συγκεκριμένα προβλήματα. Σήμερα η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ θέτει να αμφιβάλλω τις ασφάλειες αυτών των προϊόντων και είναι σε αντίθεση με πολλές γνωμοδοτήσεις εθνικών αρχών. Εγώ δεν αμφισβητώ εδώ την αρμοδιότητα και την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΦΣΑ. Αμφισβητώ το σύστημα, διότι όταν μια φυσική ουσία δεν μπορεί να αναπαραχθεί και οι αναλύσει γίνονται για συνθετικές ουσίες οι οποίες έχουν την ίδια μοριακή δομή αλλά δεν είναι οι ίδιες ε, οι οποίες είναι παρούσες στις φυσικές ουσίες είναι προφανές ε, ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δεν είναι αυτό το οποίο προστατεύει τους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, η ΕΦΣΑ συμπεριφέρθηκε έτσι σε αυτή την περίπτωση. Έκανε ανάλυση κάποιων ουσιών που είχαν την ίδια μοριακή δομή, αλλά δεν ήταν οι ίδιε ουσίε. Και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε του Ευρωπαίου πολίτε. Έτσι θέλουμε να δημιουργήσουμε τι επιστημονικέ βάσει και να προσδώσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, ή απλώ ε, διαπράττουμε μοιραία σφάλματα. Παρουσία τη ΕΦΣΑ λοιπόν και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να μου απαντήσετε συγκεκριμένα. Πρέπει να διαχειριστούμε ε, τη, ε, τον κίνδυνο της χρήσης των ουσιών, αλλά πρέπει να είμαστε και συγκεκριμένοι στις πληροφορίες μας. Διότι ελοχεύει ο κίνδυνος να τεθούν εκτός αγοράς κάποιες ουσίες και απλώς η ΕΦΣΑ να είναι ένα εργαλείο διαχείρισης της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ορισμένοι συνάδελφοι επέμειναν και είπαν ότι υπάρχει ένα διακύβευμα ακριβώς του αποτελέσματος αυτής της πρότασης σε σχέση με τις ευρωεκλογέ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν μια προστασία της υγείας τους και βλέπουμε ότι τα τρόφιμα είναι ένα στοιχείο κλειδί. Από τη μία πλευρά βλέπουμε ότι η Κομισιόν δραστηριοποιείται για να πει ότι θα αυξήσουμε τη διαφάνεια. Αλλά όταν βλέπω στο κείμενο και επίσης στις προτάσεις σας κυρία εισηγήτρια ε, θέματα τα οποία είναι οπισθοδρόμηση όταν βλέπω ότι προτείνεται να υπάρχει μια αποκάλυψη μετά την δημοσίευση ε, του καταλόγου της ΕΦΣΑ και όχι πριν. Ο στόχος είναι να υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία προτού δοθεί η επιστημονική γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Δεν συμφωνείτε πάνω σε αυτό. Όταν βλέπω πριν ή τα κράτη και η Κομισιόν είχαν πρόσβαση σε στοιχεία εμπιστευτικά, εσείς θέλετε να καταργήσετε η ΕΦΣΑ να μπορεί να αποκαλύπτει στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη εμπιστευτικές πληροφορίες. Γιατί γλύφωσα τη ζητήσαμε συμπληρωματικές μελέτες. Λέτε ότι μόνο η ΕΦΣΑ μπορεί να το ζητήσει αυτό. Όχι, θα πρέπει να είναι η Επιτροπή, θα πρέπει να είναι τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να ζητά από την ΕΦΣΑ να κάνει συμπληρωματικές μελέτες. Περιορίζεται την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Όταν μου μιλάτε για πληροφορίες εμπιστευτικές, μα ποιες εμπιστευτικές πληροφορίες όταν ζητούμε να έχουμε πρόσβαση στις μελέτες για την υγεία και το περιβάλλον, γιατί τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά ε, για τους ε, και για τους βιομήχανους. Η ΕΦΣΑ δεν μας έδωσε τις 74 μελέτες σχετικά με την αξιολόγηση της γλυφοσάτης ε, και ότι ο Οργανισμός Υγείας δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά και μας λέτε ότι είναι ιδιοκτησία ε, των βιομηχάνων, βρίσκεται ότι είναι φυσικό. Όταν ζήτησα την ΕΜΑ μου λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα το εμπιστευτικό. Αλλά επειδή φοβάται τους συνγόρους της βιομηχανίας, η βιομηχανία λέει ότι είναι εμπιστευτικά στοιχεία. Ας βάλουμε τα πράγματα επιτάπητος. Είμαστε υπέρ της ανεξαρτησίας των εμπειρογνωμόνων. Και εδώ είναι το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους που αξιολογούν τους κινδύνους και αυτούς που διαχειρίζονται τους κινδύνους. Όταν η ΕΦΣΑ ε, ζητά να δώσουμε συμβουλέ στους βιομηχανου, πολύ καλά, αλλά δεν θα πρέπει να είναι οι ίδιοι που αξιολογούν τους κινδύνους. Όταν λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ΕΦΣΑ, εγώ είμαι υπέρ, αλλά με αποδείξεις να υπάρχει πράγματι ανεξαρτησία των εμπειρογνωμένων, να δίνεται όλα τα στοιχεία και να μην κρύβεστε πίσω από την εμπιστευτικότητα για τους βιομηχάνους. Εγώ είμαι επιστήμον. Πώς μπορώ να δεχθώ επιστημονική γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ αν δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στα, στα στοιχεία βάσης. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε θα πρέπει να βάλουμε όλα τα χαρτιά επιτάπητος και να δείξουμε στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο είναι απαιτητικό και θέλουμε όλα να είναι διαφανή. Κύριε Σόμερς, είπατε τα πρωτόκολλα πρέπει να δίνονται, τα πρακτικά, να ξέρουμε ποιος ψηφίζει τι. Πολύ καλό. Ναι, είναι καλό αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα που πρέπει να βελτιωθούν στο κείμενο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ε, μας δίνουν λιγότερη διαφάνεια. Όλο και περισσότερο μιλούμε για διαφάνεια διαφάνεια, αλλά είναι ένα μέσο για να τη μειώσουμε τη διαφάνεια. Ας είμαστε απαιτητικοί απέναντι στους ψηφοφόρους μας. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Χέντεμπεργκ τώρα. Κυρία Κάντενμπαχ, ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο παρατηρήσεις πολύ θα λάβει υπόψη η συγγητριά μας. Καταρχήν μια προσωπική παρατήρηση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Όταν μιλάτε για ε, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και κάπως την αμφισβητείτε γιατί είπατε ότι έχει πάρα πολλές υπογραφές από ένα κράτος μέλος μόνο μου φαίνεται ε, ε, αξιοπερίεργο ότι αμφισβητείτε κάπως την άποψη της δημοκρατικής αυτής πρωτοβουλίας πολιτών. Όταν υπάρχουν ε, οι κανόνες του παιχνιδιού, όταν έχουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη, αυτή είναι η δημοκρατική επιταγή και αυτό οφείλουμε να το σεβαστούμε και δεν μπορούμε να το ε, ε, αμφισβητούμε. Ένα δεύτερο τώρα στοιχείο. Συμφωνώ ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, μεταξύ ε, του κλάδου, και διαφορετικές απόψεις υπάρχουν και στο Κοινοβούλιο. Ε, στην πρότασή μου, στην αγνομοδότηση που ετοίμασα για την Επιτροπή Άγκρη, εξετάζω τη δυνατότητα του νέου συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διαβουλεύσεις και των κρατών μελών αλλά θα πρέπει να είναι από, εκπρόσωποι από τον τομέα της υγείας και όχι από τον τομέα της βιομηχανίας. Ένα άλλο σημείο που αναφέρθηκε προηγουμένω εν συντομία σχετικά με τι μελέτε επαλήθευση. Το άρθρο 33ε, νομίζω ότι είναι αυτό είναι σαν να μετατοπίζεται η ευθύνη και το κόστος από τον ετούντα την άδεια προς ε, τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Αν τις ε, μελέτες αυτές πρέπει να τις κάνει η Επιτροπή, αν τον κίνδυνο πρέπει να τον διαχειρίζεται η Επιτροπή, φαντάζομαι ότι οι μελέτες αυτές θα ε, πληρώνονται και από την Επιτροπή. Και δεν είναι σαφές στην πρότασή σας ποιος θα αναλαμβάνει το κόστος ε, της μελέτης. Η παράγραφος αυτή λοιπόν ε, είτε θα πρέπει να διαγραφεί είτε ε, θα μας δώσει μια σαφέστερη εξήγηση η Επιτροπή για το πώς θα ανατίθενται αυτές οι μελέτες και ποιος θα φέρει το κόστος για την διεξαγωγή των μελετών. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια, ερωτήσεις. Αν όχι, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρούλ από την ΕΦΣΑ. Όχι. Εσείς πρώτα και μετά η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την πλευρά της ΕΦΣΑ, η πρόταση της Επιτροπής υποστηρίζει την πρωτοβουλία μας μια πρωτοβουλία που ακολουθούμε από το 2014. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι κατά τη γνώμη μας θα αποτελούσε ένα μεγάλο βήμα πρόοδου υπέρ της διαφάνειας, διότι η ΕΦΣΑ θα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να δημοσιεύει ανεπεξέργαστα δεδομένα ε, σε πολύ ευρία κλίμακα. Η ΕΦΣΑ θα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση και τους οικονομικούς πόρους να χρησιμοποιεί δομές και εργαλεία ώστε να δημοσιεύει προδραστικά ανεπεξέργαστα δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο το οποίο είναι υποσυζήτηση, αυτό το κατάλαβα αλλά δεν είναι δικό μας θέμα και κατά αυτόν τον τρόπο ακολουθούμε την προσέγγιση μας ότι τα επιστημονικά δεδομένα χρειάζονται επανεξέταση και προς αυτό χρειάζονται ακαδημαϊκοί και ερευνητές οι οποίοι πρέπει να κάνουν τους υπολογισμούς τους βάσει των ανεπεξέργαστων δεδομένων και να εξαγάγουν τα συμπεράσματά τους. Αυτό θα αποτελέσει ένα βήμα θετικό όχι μόνο για τη διαφάνεια αλλά θα δώσει και σαφήνεια στην ΕΦΣΑ για να δούμε πόσο πρέπει να προχωρήσουμε με τα θέματα δημοσιοποίησης στοιχείων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια σύγχυση, διότι μερικές φορές πρέπει να περιμένουμε να θέσει τους κανόνες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το βαθμό διαφάνειας που θα εφαρμόσουμε. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε ένα σαφές νομικό πλαίσιο, τι πρέπει να προστατεύεται και τι πρέπει να δημοσιεύεται. Κατά τη γνώμη μας, η πρόταση της Επιτροπής αυτό το καθιστά σαφές και μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να προβλέψουμε τι θα απαιτείται ε, από τους ετούντες ένα δεύτερο σημείο όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών και στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στην προεπιλογή των εμπειρογνωμόνων ε, για το πάνελ. Αυτό μπορεί να συζητηθεί για το πώς θα γίνεται στην πράξη, αλλά τα κράτη-μέλη θα μπορούν να έχουν λόγο στο διορισμό των εμπειρογνωμόνων για την ΕΦΣΑ, εφόσον η αριστεία των εμπειρογνωμόνων είναι εγγυημένη, καθώς και η ανεξαρτησία τους, σύμφωνα με την πολιτική ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ, και εφόσον εμείς στην ΕΦΣΑ μπορούμε να αποφασίσουμε για τη σύνθεση των πάνελ, δεν είναι τόσο σημαντικό για μας αν η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα γίνεται από τα κράτη-μέλη ή από την ΕΦΣΑ ή συνδυασμένα. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να έχουμε τους καλύτερους δυνατών ε, επιστήμονες που θα είναι και ανεξάρτητοι επιστήμονες. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ε, Αποζημίωση των οργανισμών στα κράτη-μέλη που μας δανείζουν τους εμπειρογνώμονες. Αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό και για τα κράτη-μέλη, γιατί αυτή τη στιγμή πρόκειται για εμπειρογνώμονες που δεν πληρώνονται από την ΕΦΣΑ και σύμφωνα με την πρόταση ε, θα υπάρχουν πόροι ώστε να αποζημιώνονται οι οργανισμοί στα κράτη-μέλη, γιατί αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να μας δώσουν τους καλύτερους. Και θα υπάρχουν και οι απαραίτητοι πόροι για να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε μπορούν να προετοιμάζουν επιστημονικό έργο για την ΕΦΣΑ. Για μας λοιπόν θεωρούμε ότι είναι σημαντικά βήματα για τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία αυτά. Υπάρχει όμως ένα αλλά. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν εφόσον υπάρχουν οι οικονομικοί πόροι. Το χειρότερο σενάριο, η χειρότερη εναλλακτική λύση θα είναι να καταλήξετε σε συμφωνία και μετά να μην υπάρχουν χρήματα στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και σα οικετεύω, μην το κάνετε αυτό, γιατί αυτό θα σημαίνει πλήρη αποτυχία. Αλλά εάν προβλεφθούν και οι κατάλληλοι πόροι, όπω προβλέπετε στην πρόταση τη Επιτροπή, η πρόταση είναι πολύ καλή για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία Τη ΕΦΣΑ και θεωρούμε θετική την πρόταση τη Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Ζόμερ για την προσπάθεια που αναγνωρίζουμε ότι έγινε σε πολύ σύντομο διάστημα η πρόταση του σχεδίου έκθεσης και μπορούμε να συζητούμε αυτή τη στιγμή και να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την πρόταση εντός ε, της ε, ε, τωρινής θητείας. Ο Επίτροπος και οι Επίτροποι Γενικών είπαν περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για την αναθεώρηση της διατροφικής νομοθεσίας και πριν κάνουμε την ε, τροποποίηση έγινε μια πολύ αναλυτική διαδικασία refit ε, της εξέτασης καταλληλότητας δηλαδή της νομοθεσίας ε, σε θέματα τροφίμων. Ζητήσαμε με πολλούς ενδιαφερομένους για μεγάλο χρονικό διάστημα και θεωρούμε ότι οι αρχές της γενικότερης νομοθεσίας για τα τρόφιμα λειτουργούν ακόμα αρκετά αποτελεσματικά και να πω ότι εμείς δεν καταλήξαμε στο συμπέρασμα ούτε αυτοί οι οποίοι ε, ε, ενδιαφέρονται για το γενικότερο διατροφική νομοθεσία ότι χρειάζεται πλήρης ε, αναδιάρθρωση και μεταρρύθμιση. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια στοχευμένη τροποποίηση. Ε, όντως εξετάσαμε και το ενδεχόμενο της πρωτοβουλίας των πολιτών για τη γλυφοσάτη αλλά σε γενικέ γραμμέ νομίζω ότι είναι προφανέ ε, σε όλου εκείνου που ασχολούνται ε, με το θέμα ε, του γενικότερου δημοσίου συμφόροντο και σίγουρα τα τρόφιμα είναι κάτι το οποίο είναι δημοσίου συμφόροντα, ότι υπάρχουν αυξανόμενε προσδοκίες από την κοινωνία, θέλουν να ξέρουν τι γίνεται στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων και πρέπει οι πολίτες να έχουν και την ευκαιρία να αντιληφθούν όσο το δυνατόν καλύτερα τι συμβαίνει. Επομένως, ε, οι δύο πτυχές ε, και όπως είπα αυτό προέρχεται και από το Refit αλλά και από τις ε, πρωτοβουλίες των πολιτών που θέλει να αντιμετωπίσει η πρόταση είναι η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματός μας, κυρίως όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων, την ΕΦΣΑ. Θέλαμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, πτυχές με φιλόδοξο τρόπο και η μεγαλύτερη διαφάνεια και όσες φορές και να το πω δεν αρκεί, ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύαμε να σχεδιάσουμε το μέσο, ο τρόπος με τον οποίο συντάχθηκε η πρόταση, έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια. Και θα πρέπει λοιπόν ε, στις περαιτέρω επαφές μας ε, να δούμε αναλυτικά γιατί κάποιοι από εσά θεωρείτε ότι είναι μικρότερη διαφάνεια από το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας και δεν αντιλαμβανόμαστε εμείς το σχεδιασμό μας έτσι. Σίγουρα ο στόχος είναι λοιπόν η μεγαλύτερη διαφάνεια και σίγουρα απαιτεί και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη νομιμοποίηση της αποστολής της ΕΦΣΑ και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη ε, στο έργο της ΕΦΣΑ και σε γενικές γραμμές θα αποτελέσει και ένδειξη ότι η ΕΦΣΑ και το σύστημα ε, είναι υπόλογο προς τους πολίτες, ε, το οποίο είναι κάτι το οποίο συμβάλλει σε ένα πιο δημοκρατικό σύστημα. Τώρα, ποιο είναι ο ακρογωνιαίος λήθος της διαφάνειας. Ο ακρογωνιαίος λήθος σε αυτή την πρόταση είναι η ε, ενεργός δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που υποστηρίζουν τις αιτήσει έγκρισης τροφίμων. Και όπως ακούστηκε, αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύτιμο εάν ε, ε, υπάρχει στην αρχή της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου, γιατί επιτρέπει στους ενδιαφερομένους, ε, στους ενδιαφερομένους πολίτες να κατανοήσουν τι ακριβώς γίνεται στη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η έγκαιρη δημοσιοποίηση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης, για να εγγυηθούμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια δημόσιο, και το δημόσιο έλεγχο. Και το έχουμε και πλαισιώσει με διάφορα άλλα στοιχεία, τη δημόσια διαβούλευση για τις μελέτες που υποβάλλονται, ε, το ενωσιακό μητρό. Όλα αυτά τα εργαλεία στόχο έχουν να εξασφαλίσουν ότι η ΕΦΣΑ θα έχει στη διάθεσή της ε, τα ευρύτερα δυνατά επιστημονικά στοιχεία ε, και επιστημονικές ενδείξεις, ώστε η ΕΦΣΑ να έχει τα καλύτερα μέσα στη διάθεσή της και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Υπήρχε μια ερώτηση και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι βέβαια το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε σε άλλη σύνθεση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να προτείνει καταλόγους, θετικούς καταλόγους πληροφοριών που θα μπορούσαν βάσει ε, δεόντως αιτιολογημένων ε, ε, ετοιμάτων του κλάδου να θεωρηθούν εμπιστευτικά. Όταν έχουμε εκατοντάδες ή και χιλιάδες σελίδες, ε, ε, επιλέξαμε να ακολουθήσουμε ένα παράδειγμα το οποίο σε πολύ καλά στον τομέα των φαρμάκων, που έγινε ακριβώς αυτό. Αν κάποιος ισχυριστεί ότι κάποιες πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι ε, εμπιστευτικές για εμπορικούς σκοπούς μόνο στους τομείς αυτούς ε, και αυτούς έχουμε συμπεριλάβει στον κατάλογο. Πουδήποτε αλλού δεν χρειάζεται να υπάρξει τέτοιο εγχειρισμό. Οτιδήποτε βρίσκεται σήμερα στους καταλόγους πληροφοριών που πρέπει να ε, είναι δημόσια διαθέσιμες καλύπτονται. Αυτό θα συνεχίσει λοιπόν να ισχύει και θα είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες. Πρόκειται για μια πρακτική προσέγγιση ώστε να μπορέσουμε να επικεντρώσουμε τη συζήτηση μόνο σε αυτούς τους τομείς. Και ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, αυτοί που ισχυρίζονται ότι το τάδε, για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι εμπιστευτικό, θα πρέπει να το αιτιολογήσουν δεόντως και να εξηγήσουν ότι αυτό θα είναι εις βάρος ε, της ε, επιχείρησής τους ε, εάν δημοσιοποιηθεί. Να πω βεβαίω ότι τίποτα σε αυτή την πρόταση δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα των πολιτών ή οποιοδήποτε άλλο για την πρόσβαση σε ε, πληροφορίες και τη σχετική νομοθεσία, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και για το ε, κυρίαρχο δημόσιο συμφέρον. Αυτά μένουν ανέπαφα. Ανέπαφα επίσης παραμένουν και τα δικαιώματα της σύμβασης του άρχους. σε καμία περίπτωση και τουλάχιστον όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς δεν πλήττεται η σύμβαση του άρχους. Ε, έχουμε δει τα όσα προβλέπονται και ε, σκοπεύουμε να παραμείνουν ως έχουν για τη σύμβαση του άρχους. Θέλω λοιπόν να είμαι βέβαιη ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως ποια είναι η πρόθεσή μας και ποιο ήταν και το γράμμα της πρότασης. Ε, πράγματι ε, ε, ουσιαστικά κάνουμε άσκηση ισορροπίας ε, και θέλουμε και ο κλάδος να γνωρίζει και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους, διότι είναι πολύ δαπανηρές αυτές οι επενδύσεις και όλοι θέλουν να προστατεύονται και τα στοιχεία τους και τα δικαιώματά τους. Και θέλω να εξασφαλίσω και σε όλους εδώ στην Ομίγυρη ότι τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα της αποκλειστικότητας των δεδομένων και φυσικά και η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων προστατεύονται. Δεν ε, υπάρχει καμία παραβίαση σε αυτή την περίπτωση. Στη συζήτηση ακούστηκε και γιατί δεν εξηγείται περισσότερο πόσο ακριβώς θα γίνει αυτό. Υπάρχει μια διάταξη στην πρόταση ότι η πρακτική εφαρμογή θα είναι αρμοδιότητα της ΕΦΣΑ και εξηγούνται και οι προϋποθέσεις και οι προϋποθέσεις είναι τέτοιες που επιτρέπουν ε, σε αυτές τις διατάξεις τις οποίες σας ανέφερα να προστατεύονται κατά την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας. Επομένως, όσοι επιθυμούν πρόσβαση στις πληροφορίες θα πρέπει να σέβονται τα όρια αυτά. Τώρα, στη συνέχεια, η πρόταση Προσφέρει επίση και τη δυνατότητα στην ΕΦΣΑ να βοηθήσει τους ετούντε ε, με συνεδριάσεις ε, πρώτη υποβολής ε, των στοιχείων τους. Θα υπάρχει και βοήθεια πρώτη υποβολής και φυσικά θα πρέπει να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της ΕΦΣΑ δεν θεωρούμε ότι η ΕΦΣΑ θα πρέπει να είναι ε, συντάκτης μαζί με τους, ε, ε, αυτούς που υποβάλλουν την πρόταση την πρόταση, της πρότασης, αλλά υπήρχε αίτηση, τουλάχιστον από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες τουλάχιστον σε αυτό και πιστεύουμε το ποιο συνάντησε ποιον ε, και τι συζήτησε σε αυτές τις ε, ε συμβουλές οι οποίες δίνονται πρώτη υποβολή, θα πρέπει να είναι γνωστό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τι ε, μελέτες επαλήθευση. όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή η ΕΦΣΑ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επιστημονικές μελέτες οι οποίε είναι απαραίτητε για την ε, εκπλήρωση τη αποστολή τη. Αυτά μένουν ως έχουν, δεν αλλάζουν, αλλά Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρετικές περιστάσεις, ε, ιδίως όταν κάποιο θέμα είναι ιδιαίτερα επίμαχο βάσει των οποίων να χρειάζονται κάποιε εξασφαλίσει ότι ελήφθη υπόψη η καλύτερη δυνατή επιστημονική ε, γνωμοδότηση. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από την ΕΦΣΑ να ζητήσει επιπλέον μελέτες ε, για σκοπούς επαλήθευση. Εμεί θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, το οποίο θα μείνει στην αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη συνοχή. Ρωτήθηκε πώ θα χρηματοδοτηθεί αυτό. Ε, περιλαμβάνεται στην πρόταση ως κάτι το οποίο χρηματοδοτείται από δημόσια κονδύλια. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το δημόσιο πληρώνει ε, για τις ε, αιτήσει του κλάδου είναι για πάρα πολύ συγκεκριμένα επιστημονικά κενά τα οποία μπορεί να ανακύψουν ε, σε κάποια περίπτωση και πραγματικά πιστεύω σε εξαιρετικές περιστάσεις και μόνο. Υπάρχει λοιπόν δημόσιο συμφέρον να συμπληρωθούν αυτά τα κενά με αυτές τις μελέτες επαλήθευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί επίσης πάρα πολύ σημαντικό ε, το να συμμετέχουν περισσότερα κράτη-μέλη στην ε, Ευρωπαϊκή Επιρογνωμοσύνη. Εδώ πρόκειται για τη βιωσιμότητα του συστήματος. Η πρόταση να συμμετέχει ο εκτελεστικό διευθυντή ε, τη ΕΦΣΑ. Ε, ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο τη ΕΦΣΑ ποια είναι τα βασικά κριτήρια τα οποία είναι απαραίτητα για την επιλογή των εμπειρογνωμόνων, ιδίω όταν ε, μα ενδιαφέρει η αριστεία, η ανεξαρτησία και η καλύτερη δυνατή σύνθεση ενό πάνελ ο εκτελεστικός διευθυντής ε, μπορεί κάλλιστα να ε, ζητήσει να υπάρξει πρόσκληση ενδιαφέροντος ε, από εμπειρογνώμονες, όπως γίνεται και σε άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες, για να έχει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν υπήρξαν αρκετά αιτήματα για την αύξηση της διαφάνειας, όχι μόνο στη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου, αλλά και της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου. Και εδώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει ξεχωριστή πρόταση που ε, τροποποιεί τον κανονισμό της επιτροπολογίας προς αυτή την κατεύθυνση, ιδίως όσον αφορά την ε, συμμετοχή της Επιτροπής Υποβολής ε, Ενστάσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται αυτή τη στιγμή ε, στο Συμβούλιο. Επίσης, η πρόταση θέτει τα θεμόλια για να υπάρχει μια συνολική ε, στρατηγική επικοινωνίας κινδύνου. Αυτά είναι πέραν της ΕΦΣΑ, είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη που πρέπει να συμμετέχουν στη στρατηγική. Πολύ συχνά αυτό που θεωρείται έλλειψη διαφάνειας στη διαχείριση κινδύνου είναι στην πραγματικότητα μια ένδειξη ε, επικοινωνίας ε, που δεν είναι αρκετά αποτελεσματική για να ε, διαβιβάσουμε ποιος ακριβώς είναι ο κίνδυνος. Επομένως, θέλουμε να έχουμε επικοινωνία του κινδύνου όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσον αφορά τον προπολογισμό και του πόρους, ε, νομίζω ότι είναι σχεδόν αυτονόητο αυτό. Ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα θα έχει κάποιο κόστο ε, και ο προπολογισμό και οι πόροι έχουν ε, προβλεφθεί. Έχουν προβλεφθεί τα στοιχεία. Ο προπολογισμό ακόμα δεν έχει εγκριθεί, αλλά... Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε την πρόταση χωρίς να υπάρχουν και κατάλληλοι πόροι στον προπολογισμό. Η πρόεδρος προτρέπει την ομιλήτρια να ολοκληρώσει. Ναι. Να σας πω κάτι τελευταίο όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της νομοθετικής πρότασης και της ε, αρμόδιας επιτροπής. Είναι δέσμευση του Επιτρόπου μας ε, που την έχει κάνει επανειλημμένος τα αποτελέσματα της Επιτροπής για τα φυτοφάρμακα ε, και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αρκετές πρωτοβουλίες, ε, ε, εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίες για συγκεκριμένους ουσίες και προϊόντα, θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία που είναι σε εξέταση, που είναι το refit της νομοθεσίας φυτογενομικής προστασίας. Δεν παρεμβαίνουμε στο έργο της Επιτροπής Φυτοφαρμάκων, ίσα ίσα περιμένουμε τα αποτελέσματα γιατί ε, είναι και η κατάλληλη στιγμή να τα λάβουμε υπόψη στη διαδικασία του ρηφή των φυτογεωνομικών προϊόντων. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και την εισηγήτρια και όλους για τη δυνατότητα αυτή ανταλλαγής απόψεως. Η κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να είχα ακούσει από την Επιτροπή και κάτι για τη σύμβαση του Όρχους. Γιατί και σε άλλες επιτροπές έχει αναφερθεί. Ίσως η Επιτροπή μπορεί να μας δώσει τις πληροφορίες αυτές εκ των υστέρων. Ευχαριστώ πολύ όλους για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σημείωσα πολλά ε, ενδιαφέροντα και περιμένω τις τροπολογίες που θα υποβληθούν. Είμαι σχετικά αισιόδοξη ότι μπορεί να τα καταφέρουμε. Είμαι πιο αισιόδοξη τώρα από ό,τι στην αρχή αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση αυτή. Η ημερομηνία για υποβολή των, τροπολογιών είναι 11 Σεπτεμβρίου και ε, στην Ένβη Επιτροπή 12 Νοεμβρίου η ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. 14η συνεδρίαση των μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, COP14. Εξετάζουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος. Έχουμε ε, συνεισηγητές ή και κάποιους που αντικαθιστούν τους εισηγητές. Για τον κύριο Λίνς η κυρία Κόνι Λάκεν. Κυρία Πρόεδρε, εκπροσωπώ εδώ τον κύριο Νόρμπερτ Λίντς που είναι συνεισηγητής. Η COP14 υπάρχει εδώ και χρόνια και μάλιστα εορτάζουμε και την επέτειό τη και δείχνει πόσο σημαντικό είναι να καλύπτουμε τα θέματα αυτά της βιολογικής ποικιλότητα. Όλοι οι συνάδελφοι θεωρούμε απαραίτητο να ενταθούν οι προσπάθειες για την βιοποικιλότητα ώστε στη μελλοντική περίοδο να είναι ακόμη πιο ε, εντατικές οι προσπάθειες σε σχέση με την περίοδο 2011-2020 με πιο φιλόδοξες στρατηγικές για την περίοδο μετά το 2020 καθώς ε, και χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό υλοποίησης ε, όταν εργαζόμαστε με την προοπτική του 2050. Σε ένα ψήφισμα λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, ζητάμε να λαμβάνει υπόψη την βιοπικιλότητα όχι μόνο τους δικούς μας στόχους, αλλά και τους παγκόσμιους στόχους για το 2020. Τώρα για τη στρατηγική και το όραμα για το 2050 ε, θα συζητηθεί ε, στην COP14 ε, στην Αίγυπτο θα πρέπει να συμβαδίζει με την, το θεματολόγιο το 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη και τους περαιτέρω στόχους. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, να εντείνουμε τις προσπάθειες για την υλοποίηση των στόχων του 2020, να εντείνουμε τις προσπάθειες για ε, την περίοδο μετά το 2020 και να δοθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση. Στο ψήφισμά μας αναφέρουμε έξι σημεία και θα ήθελα τα δύο από αυτά να τα αναφέρω συγκεκριμένα. Καταρχήν, ζητάμε ένα ισχυρό διεθνές ε, πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020 και θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένο να έχουμε βασικούς δείκτες ε, προόδου για να μπορούμε να παρακολουθούμε την υλοποίηση και την προστασία της βιοπικιλότητας. Αυτά είναι σημαντικά θεμαία για να μπορέσει να λειτουργήσει η στρατηγική μας για το όραμα του 2050 για τη βιολογική ποικιλότητα. Και παράλληλα θέλω να τονίσω ότι είναι σημαντικό να είμαστε ρεαλιστικοί, να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις και να μην υπερβαίνουμε αυτά τα οποία είχαν ε, ήδη προσδιοριστεί στο Παρίσι. Δεύτερον, οι θετικές συνεισφορέ ε, της ε, δασοκομεία και της γεωργία για τη βιοπικιλότητα σχετίζονται άμεσα και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να φροντίσουμε, να υποστηρίζουμε τις ορθές γεωργικές πρακτικές για να εξασφαλίσουμε τα οικοσυστήματα και τα διάφορα είδη. Ζητάμε λοιπόν από τους εταίρους να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπάλας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε θέμα της βιοπικιλότητας ανεβαίνει στη συνείδηση των συμπολιτών μας και μπορούμε να πούμε ότι ήταν μέρος μιας πολιτικής κρίσης στη χώρα μου εδώ και δύο μέρες εφόσον ο Υπουργός Οικολογίας παρετήθηκε λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει καθόλου δράση από πλευράς της κυβέρνησης της Γαλλικής και σε επίπεδο διεθνές και ευρωπαϊκό που οδήγησε σε μείωση 80% του αριθμού των πτηνών και εντόμων. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε μια στιγμή, εδώ ε, έχουμε λιγότερο από ένα χρόνο για τις ευρωεκλογέ, όπου η συνείδηση των συμπολιτών μας αφυπνίζεται για ένα θέμα που δεν τους άγγιζε πριν από λίγο καιρό. Είναι λοιπόν σημαντικό σήμερα να δράσουμε και από την άποψη αυτή καταβάλλονται προσπάθειες και είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε και να παρατηρήσουμε. Για να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, ε, είμαι αρκετά ευτυχής που οι περισσότεροι είναι αυτής της άποψης. Υπάρχουν βεβαίως συμφέροντα, νόμιμα ε, και βεβαίως ως προς την απασχόληση στην ενεργεία μπορεί να οδηγήσει σε επιφυλάξεις. Ε, πρέπει να εντάξουμε στο σύνολο των ε, πολιτικών μας την βιοπικιλότητα. Δεν είναι ένας ε, τομέας, είναι μια προσέγγιση, μια προσέγγιση πολυκλαδική κατά κάποιο τρόπο και θα κλείσω λέγοντας ότι υπάρχει ένα στοιχείο σημαντικά. νομίζω ότι πολύ συχνά ε, η ΚΟΠ είναι σημαντικά, σημαντικές στιγμές, αλλά πολύ συχνά δεν ακολουθούνται από πράξεις και καμιά φορά υπάρχει και ο σε ορισμένους τομείς και από την άποψη αυτή μπορούμε να είμαστε κάπως ανήσυχοι μετά την υπογραφή ε, των στόχων IC. Δεν έχουμε πραγματική αξιολόγηση για να δούμε πού βρισκόμαστε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν δείκτες σήμερα ούτω ώστε να μπορέσουμε ε, να αξιολογήσουμε ε, τις πολιτικές μας ή θα έχουμε δομές που δεν θα μπορούμε να αξιολογήσουμε και δεν θα ξέρουμε αν αυτό που κάνουμε είναι αποτελεσματικό είναι αυτό σημαντικό, αλλά για τα υπόλοιπα αυτή η συνειδητοποίηση συνολική θα πρέπει να διευρυνθεί και νομίζω ότι η εργασία πάει προς την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πουστέκ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι η διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα και ε, στην Πολωνία ε, αυτή είναι η περίπτωση το 2015 εφαρμόζοντας ε, την σύμβαση ένα ειδικό πρόγραμμα προστασίας της βιοπικιλότητας και της αηφορίας υιοθετήθηκε με ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης 2015-2020 νέο πλαίσιο και νέα στρατηγική μετά το 2020 για την διατήρηση της βιοπικιλότητας θα πρέπει να είναι κάτι το φίλο. Είναι προφανές η προκαταρκτική εργασία θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους με την συμπερίληψη των ενδιαφερομένων ενώσεων, οργανώσεων, επιχειρήσεων και άλλους. Η διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και ε, στην παγκόσμια αξιολόγηση και να μεταφράζεται στην εφαρμογή ε, της επίτευξης των στόχων της σύμβασης Στην νέα στρατηγική στόχη για την διατήρηση της βιοπικιλότητας θα πρέπει να έχουν δείκτες μετρήσιμους και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι νέοι στόχοι βασίζονται σε βιώσιμους στόχους ανάπτυξης και ότι έχουν προστιθέμενη αξία για την εφαρμογή των στόχων ε, των, της ε, σύμβασης. Περιλαμβάνεται και η βιοπικιλότητα σε πάρα πολλούς τομείς. Ενέργεια, ορυχία, υποδομές, παραγωγή, ε, μεταποίηση και υγεία η βιοπικιλότητα πρέπει να είναι μέρος όλων αυτών των τομέων. Θα πρέπει επίσης να εστιαστούμε ε, στην ύπαρξη στενοτέρων δεσμών ανάμεσα στην βιοπικιλότητα και στην κλιματική αλλαγή. Τα δύο αυτά πράγματα θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα αλληλένδετο πράγμα. Έχουμε την κλιματική αλλαγή που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για την βιοπικιλότητα, ενώ από την άλλη πλευρά μια καλή σύμβαση θα μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε ε, και να παρεμποδίσουμε με την αρνητική κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Η βιοπικιλότητα είναι κάτι το οποίο γίνεται αυξανόμενο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κατάσταση επιδεινώνεται όλο και περισσότερο και πρέπει να κάνουμε κάτι. Και πάντοτε αυτά γίνονται. Ε, ό,τι γίνεται είναι εις βάρος της βιοπικιλότητας, της χλωρίδας, της ε, πανίδας, ε, της κτηνοτροφίας, όχι μόνο εδώ στην Ευρώπη αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. η κτηνοτροφία αυτή την ε, εποχή έχει αρνητικές επιπτώσεις ε, στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στην Οκεανία σχετικά με τις ζωοτροφές και το είδωρ 20% χρησιμοποιείται για την κτηνοτροφία και οδηγεί σε λήψεις ε, ύδατος, ε, σε αέρια και δημιουργεί πάρα πολλά άλλα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σχέδιο δράσης συνολικό, περιεκτικό, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βιοπικιλότητας και να μην ξεχνούμε και την κτηνοτροφία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έκλεισε ο κατάλογος ε, των ε, ομιλητών. Η κυρία Λουντού από την Κομισιό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρα. Θα ήθελα εκ μέρου Κομισιόν ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το καλό σχέδιο ψηφίσματος και την υποστήριξη σας ε, για την COP14. Συμφωνούμε με πολλά σημεία αυτού του σχέδιου ψηφίσματος. Συμφωνούμε ότι μας ανησυχεί ότι ε, σχετικά με τους στόχους IG υπάρχει κάποια καθυστέρηση και έχουμε κακή κατάσταση ε, στην COP15 ε, θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία ε, για το συνολικό παγκόσμιο πλαίσιο βιοπικιλότητας μετά το 2020 σχετικά με τις δεσμεύσεις στην εφαρμογή. Όπως γνωρίζετε, ετοιμάζουμε με τα κράτη-μέλη για τα συμπεράσματα για την COP15 και όπως ζητήθηκε από την όλη διαδικασία, εμείς και τα κράτη-μέλη ε, την περασμένη εβδομάδα έχουμε ανταλλάξει απόψεις και υποβάλει ε, στον γραμματέα ε, μερικές απόψεις και αναφέρουμε ότι η διαδικασία θα πρέπει να επιτρέψει την ανάπτυξη ρεαλιστικών, φιλόδοξων και εφικτών μετρήσιμων στόχων για να ενισχύσουμε κατάσταση. Το πλαίσιο θα πρέπει επίσης να προβλέψει συμπληρωματικούς μηχανισμούς ε, και επίσης εθελοντικές δεσμεύσεις ε, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της βιοποικιλότητας που να προέρχονται από κράτη και ενδιαφερόμενους. Θα πρέπει η διαδικασία να είναι διαφανής, πλήρης και νομίζω ότι συμφωνούμε με το σχέδιο ψηφίσματος και περιμένουμε την συνεχή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συζήτηση. Τώρα, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 5 Σεπτεμβρίου, 11 η ώρα και ψηφοφορία 10 και 11 Οκτωβρίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Εδώ έχουμε κοινή συζήτηση για την ε, πρόταση κανονισμού και απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος ορίζων ε, Ευρώπη. Πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Θα τα δούμε από κοινού τα δύο σημεία αυτά. Εξετάζουμε τα σχέδια γνωμοδότησης και θα ξεκινήσουμε με τον εισηγητή, τον κύριο Μπουσόη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Horizon Ευρώπη θα είναι το ένατο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας ε, και έχει 13 ε, εκατομμύρια παραπάνω από το Horizon 2020 και είναι και το πιο φιλόδεξο πρόγραμμα που έχουμε μέχρι σήμερα και γι' αυτό πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από τις προηγούμενες επιτυχίες και τα διδάγματα των προηγούμενων προγραμμάτων, το Ορίζοντας Ευρώπη θα προσπαθήσει να ενισχύσει την επιστημονική βάση της Ένωσης, να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα και να προσπαθήσει να έχει σημαντικό ρόλο στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Από την υπερθέρμανση του πλανήτη, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία. Το ορίζοντας 2020, για παράδειγμα, είχε επιτυχία διότι κατάφερε να έχει εξαιρετική έρευνα, όπως αποδείχθηκε από τις πολλές αναφορές που έχουμε σε ε, επιστημονική βιβλιογραφία για τις δημοσίευσεις του ορίζοντα 2020, αλλά το οικοσύστημα ακόμα δεν βοηθά ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε σε καινοτομία που θα έχει απτά και ε, σημαντικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός αυτών των προγραμμάτων κατά την άποψή μας ακόμα παρακολύεται από κάποιες ε, ε, σύνθετες διαδικασίες που δεν επιτρέπουν να έχουμε ταχύτερη καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνέχεια του προγράμματος πλαίσια θα βοηθήσει να έχουμε απλοποίηση και να ενισχύσουμε και το εμπορικό σήμα του ορίζοντα. Ε, όπως ε, είπε και η πρόεδρος, έχουμε κοινή συζήτηση, επομένως θα κάνουμε παρατηρήσεις και για την άλλη γνωμοδότηση. Ε, μου αρέσει η δομή των τριών πληρώνων. Ο πρώτος είναι η ανοιχτή ε, επιστήμη, οι ε, προκλήσεις και η καινοτομία στη συνέχεια και υπάρχει και το Ερευνητικό Συμβούλιο οι δράσεις ε, Μαρή Κορδόφσκα Κιουρί και το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Επίσης, καλωσορίζω τη συνέχεια των ενισχύσεων ως ε, το βασικό μοντέλο χρηματοδότησης για τον ορίζοντα Ευρώπη. Ε, το νέο πρόγραμμα βέβαια έχει κάποιες ελλείψεις οι οποίες έχουν ε, διαπιστωθεί και από την εξωτερική και από την εσωτερική αξιολόγηση και το διάλογο με τους νομοθέτες και τους ενδιαφερομένους. Και χαίρομαι και για τον αριθμό των νέων στοιχείων που έχουμε στο νέο ορίζοντα Ευρώπη ε, το οποίο θα ενισχύσει τα προγράμματα, όπω η έννοια των αποστολών, που κατά την άποψή μου θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω και γι' αυτό επέβαλα και τι τροπολογίε 10 και 11 στον κανονισμό. Όσον αφορά τη δομή του προγράμματο, υπάρχει μείωση στον αριθμό των ε, θεμάτων που είχαμε σε σχέση με τον ορίζοντα 2020 και η αναφορά στο περιβάλλον δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη δομή που έχουμε σε κλάστερ. Ε, αναφέρεται κάπου στον τομέα της υγείας, αλλά είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ε, οι ε, ε, πολίτες, χρόνιες, παθήσεις κλπ. Θέλουμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό και για τον ορίζοντα Ευρώπη και για τον τομέα της υγείας. Τώρα, η διανομή των κονδυλίων ε, δεν ε, αρκεί για να βοηθήσουμε κάποιους τομείς. Ε, στην τροπολογίες μου 20 και 23 λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει η ίδια αρχή της αναλογικότητας όπως είχαμε στον ορίζοντα 2020 το 70% θα πρέπει να εστιάζει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κοινωνίας και στη βοήθεια της κοινωνίας και το υπόλοιπο 30% θα πρέπει να εστιάζει στην βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Όσον αφορά τις αποστολές, ε, στη γνωμοδότησή μου προτείνονται κάποιες ε, ε, σημαντικές αποστολές με μεγάλο αντίκτυπο για την κοινωνία που θα βοηθήσει να συμμετέχει η επιστημονική και η επιχειρηματική κοινότητα και να αποτελέσει και καταλήτη για τους πολίτες. Ο καρκίνος είναι μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και επειδή το 70% των Ευρωπαίων θέλουν να κάνει περισσότερη Ευρώπη στον τομέα της υγείας, θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό ως προτεραιότητα στον τομέα της έρευνας. Άλλωστε, ο καρκίνος εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη μορφή θανάτου ε, στα παιδιά και η έρευνα είναι κατακαιρματισμένη στον τομέα αυτό. Επομένως, ε, δεν μπορούμε να επιτύχουμε βιώσιμα αποτελέσματα ε, απευθεία. Προτείνω λοιπόν στην τροπολογία 7 μία πρώτη ε, έρευνα για την υψηλή θνησιμότητα ε, και να μειώσουμε τον παιδιατρικό ε, καρκίνο μέχρι το 2030. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Από τον πυλώνα 2, τρεις από τους πέντε τομείς ε, έχουν άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Περιβάλλοντος και καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της χρηματοδότησης του πυλώνα 2, 32,7 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Οι άλλοι πυλώνες ε, και τομείς καλύπτουν τομείς οι οποίοι είτε άμεσα είτε άμεσα σχετίζονται με τις εργασίες του, της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είπα ότι το μέσο υγεία δεν είναι αναλογικό με τι προσδοκίε των πολιτών μα και όσον αφορά τον ε, ε, κατανομή των προπολογισμού, να επενθυμίσω τι τροπολογίε 13 και 14, ώστε να έχουμε τουλάχιστον τον ίδιο προπολογισμό με τον ορίζοντα 2020, ε, να είναι το 7% ε, και όχι το 17% και όχι το 8,1% όπως προτείνεται και από το παράρτημα 1 θα θέλαμε να περάσουμε κάποια στοιχεία από τον τομέα της υγείας να πάνε στον τομέα της ε, ψηφιακής βιομηχανίας. Αυτές είναι οι τροπολογίες 26 και 35. Τέλος, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, έχω καταθέσει αρκετές τροπολογίες για τα θέματα αυτά στην απόφαση 38, 39, 40, 41, 43, 46 μέχρι και 51 για να έχουμε καθαρές ε, λύσεις, ε, μείωση της χρήσης του άνθρακα, προστασία του αρκτικού οικοσυστήματος, μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων και μείωση των ε, ποσοστών θνησιμότητας για τους επικονιαστές. Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για προτάσεις και συζητήσεις από τους υπόλοιπους συναδέλφους και τους κοιόδης συγητές και ε, προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σα ε, για να βελτιώσουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι πολύ καλή κατά την απόψή μου αλλά θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο αποτελεσματική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και στρέφομαι στου σκιώδεις εισηγητές ή όσους αντικαθιστούν τους σκιώδεις εισηγητές όπως η οσου αντικαθιστουν του σκιωδεις εισηγητες οπω η κυρια καβεζον που της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον συνάδελφο Τίμο Βόλκεν, ο οποίος δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Μπουσόη. Με, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό μετά όσα προτείνει. Εξετάζουμε και τη συμβολή και των άλλων εισηγητών και ο αρμόδιο επί της ουσίας εισηγητή του στην Ήτρα και πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν χρειάζεται δεν να σας υπενθυμίσω ότι αυτό μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπίσουμε και τις κοινωνικές προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε προσπάθεια να αυξήσει τον προπολογισμό, αλλά αν λάβουμε υπόψη και την αύξηση των τιμών, είναι ανεπαρκής αυτή η αύξηση και ε, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προκλήσεις, αλλά και το γεγονός μου ότι ένα στα τέσσερα προγράμματα, όσο καλό και αν είναι, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα. Επομένως, χάνονται πολλές ευκαιρίες, πρέπει να αυξηθεί ο προπολογισμό στα 120 δις. Ε, η δομή όντω διατηρεί τους τρεις πυλώνες και δίνει έτσι και τη δυνατότητα προβλέψεων, αλλά υπάρχουν και σημαντικές αλλαγές που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Οι βασικοί πυλώνες, κυρίως ο πυλώνας 2, δεν έχουν τόσες πολλές λεπτομέρειες και δεν αναφέρονται σε κάθε θεματολογία συγκεκριμένα και θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ανταγωνιστική οι μεταξύ τους όσον αφορά τη χρηματοδότηση και κάποια από αυτά τα θέματα μπορεί τελικά να μην χρηματοδοτηθούν ε, ενώ θα έπρεπε. Θα πρέπει λοιπόν τουλάχιστον σε κάποια προγράμματα να υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση πιο αναλυτική. Επίσης, εδώ συμφωνώ με το συντάκτη της νομοδότησης, οι κοινωνικές προκλήσεις με τη βιομηχανία μπορεί να, ε, έτσι όπως αναμειχνύονται, μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση και δεν θα πρέπει να τα προχωρήσουμε έτσι. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το ποσοστό. Η καινοτομία είναι πολύ σημαντικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και το μεγάλο κενό και πρέπει να την προωθήσουμε, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι σημαντικό και να συμμετέχει ο κλάδος και ε, να γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στο ορίζοντα 2020 δεν θα πρέπει να μειωθεί ε, σε καμία περίπτωση γιατί είναι ο βασικός ε, τομέας ο οποίος βοηθά ε, την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αριστεία παντού και να υπάρχει και μεγαλύτερο αριθμό περιφερειών που συμμετέχουν στα προγράμματα. Θα πρέπει να βρεθεί ένα μηχανισμό ώστε η αξιολόγηση να πρημοδοτεί τα προγράμματα και όχι ε, να ε, τροφοδοτούνται μόνο συγκεκριμένε περιφέρειες, να μπορούμε να εφαρμόσουμε προγράμματα για να επιστρέψουν τα ταλέντα σε περιοχέ στις οποίες λόγω διαφορών, ε, διαφορών δυσκολιών αποχώρησαν και ε, να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να διατηρήσουμε τα ταλέντα και να αυξήσουμε την αριστεία και θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι δείκτες οι οποίες θα επιτρέπουν να αυξήσουμε, όπως είπα, την αριστεία. Όσον αφορά τι συγκεκριμένε προκλήσει, τα κλάστερ από πλευρά ε, Επιτροπή Περιβάλλοντο, σίγουρα ε, μα ενδιαφέρουν τα θέματα τη υγεία και του κλίματο. Λίγο πιο σιγά ε, να μιλάει ο μιλήτρια, λέει η πρόεδρος. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν θέματα που είναι αρμοδιότητα της έμβια, αλλά όπως είπε και ο συντάκτης ε, της νομοδότησης, η υγεία θα πρέπει να την χάνει μεγαλύτερη μεριδίου. Ε, ο καρκίνος είναι πολύ σημαντικό, αλλά και οι καρδιακές παθήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ανισότητες στον τομέα της υγείας και επομένως θα πρέπει να υπάρχει ε, και κατάλληλη χρηματοδότηση. Σίγουρα ο παιδικός καρκίνος και γενικότερα οι παιδιατρικές παθήσεις και φυσικά η μικροβιακή εντοχή. Δεν θα ήθελα βεβαίω εδώ να ξεχάσουμε και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε το περιβάλλον και να υπάρχει και συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό. Και επίση πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή η γεωργία στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι θα περιοριστεί και επομένω ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια βιώσιμη γεωργία και να. Ε, λαμβάνουμε υπόψη και τι πρόκληση αποτελεί αυτό και να υπάρχει σχετική χρηματοδότηση. Τέλος, να πούμε ότι δεν είναι τα πάντα μόνο τεχνολογία. Πρέπει να υπάρχει και σαφή ένταξη της κοινωνικής ε, ε, επιστήμης και της ανθρωπολογίας. Πρέπει να σταθούμε κυρίως στο θέμα της μετανάστευσης εδώ. Εδώ η επιστημονική διπλωματία θα πρέπει να έχει ε, μεγαλύτερο αντίκτυπο. Και τέλος, όσον αφορά τον αντίκτυπο, πολλές φορές μετράμε το πρόγραμμα της επιστημονικής έρευνας με χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει να δούμε και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Η επιστήμη ε, πρέπει να δώσει απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες ανισότητες. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς έχουμε πρόσβαση στα αποτελέσματα. Όχι μόνο την απόκτηση των αποτελεσμάτων, αλλά πώς επωφελούνται οι πολίτες από αυτά τα αποτελέσματα. Τέλος, ε, τα θέματα φύλου. Τα θέματα φύλου σίγουρα πρέπει να ληφθούν υπόψη και πρέπει να μελετηθεί και ο αντίκτυπος των θεμάτων φύλου. Και χρειαζόμαστε και τέτοια πράγματα ε, στον τομέα τομέα του φύλου και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τη συμμετοχή των γυναικών και το ποσοστό των γυναικών ερευνητών και επικεφαλής προγραμμάτων. Ε, καλό πρόγραμμα, καλή πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία μπορούμε να βελτιώσουμε και να συγχαρώ τον κύριο Μπουσάη για τη γνωμοδότησή του, γιατί πιστεύω ότι οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Now... Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μάθιες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που ξανά είμαι κοντά σας στην Επιτροπή αυτή. Το ECR γενικά συμφωνεί με την ε, κατεύθυνση της πρότασης της Επιτροπής για τα θέματα που συζητάμε. Βέβαια, όπως πάντοτε, έχουμε κάποιες ε, κριτικές παρατηρήσεις, γιατί κάθε πρόταση θέλουμε να ξέρουμε αν δίνει άριστη, ε, άριστα επιστημονικά στοιχεία, αν είναι διαφανής και αν είναι αποδοτικές για τους ε, καταναλωτές. Δεν θα λάβουμε υπόψη εθνικές προτεραιότητες και χρηματοδοτήσεις, αλλά θα επικεντρωθούμε στα θέματα όπου η διεθνής ε, προσπάθεια μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα από ότι οι εθνικές ή περιφερειακές προσπάθειες και θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία συμπληρώνοντας τις επενδύσεις που γίνονται σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό, συγγνώμη, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ο στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη με τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν όλα τα επίπεδα επιχειρήσεων και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποφεληθούν. Ως ε, Βρετανός ε, Ευρωβουλευτής ε, γνωρίζω ότι η Βρετανία δεν θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο όπως ε, και όλα τα άλλα θέματα σε σχέση με το Brexit. Όλα αυτά είναι στα χέρια των διαπραγματευτών και δεν ξέρουμε ακριβώς ε, πώς θα έχει το μέλλον. Πολλοί όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελαν να έχουμε κάποιο είδους συμμετοχή στο πρόγραμμα Horizon και αν αυτό καταστεί δυνατόν η διεθνή επιστημονική συνεργασία που ίσχυε και πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που πολλές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη έχουν με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό θα ήταν να συνεχιστεί. Τέλος, θέλουμε να έχουμε μια ισορροπία στα μέσα που χρησιμοποιούνται για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους αποδέκτες. Θέλουμε να έχουμε τους καλύτερους επιστήμονες και τα καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. κυρία Ρίης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον ε, κύριο Μπουσόη στα περισσότερα θέματα τα οποία ανέφερε και σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής. Η βασική προτεραιότητα ε, είναι να ε, είναι εγγυημένη η συνέχεια με το τωρινό πλαίσιο Horizon 2020. Επομένως, ε, το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα, το πρόγραμμα να έχει συνέχεια που θα είναι θετική για την διαφάνεια και για τους ερευνητές. Οπότε θέλουμε σωστά κριτήρια για την επιλογή των προγραμμάτων, να υπάρχει, ε, να υπάρχουν κατάλληλοι πόροι ε, και εφόσον ο πυλώνας για την υγεία είναι ένας από τους πυλώνες που πρέπει να έχει ιδιαίτερη σημασία, θα πρέπει να της δοθεί ιδιαίτερη σημασία και αντίστοιχη χρηματοδότηση θα θέλουμε να ε, μειώσουμε το διοικητικό φόρτο. Όλοι οι ερευνητές μας λένε ότι θέλουν να μειωθεί η γραφειοκρατία, να έχουμε απλουστευμένες διαδικασίες και να διασφαλίζουμε καλύτερες συνέργειες και συνεργασία με τα άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα αποδώσει καλύτερα και επί της ουσίας και ε, τυπικά, διότι το Horizon Ευρώπη θα χρηματοδοτεί ε, προγράμματα τα οποία έχουν εγγυημένη απόδοση. Παράλληλα με την ε, διάχυση των αποτελεσμάτων που θα είναι μια ε, ε, συνθήκη που θα υπάρχει ήδη στη σύμβαση με τους ερευνητές και εφόσον θα επικεντρωνόμαστε στα στοχευόμενα αποτελέσματα. Αυτή είναι μια λογική την οποία θα πρέπει να υλοποιήσουμε, να ενθαρρύνουμε και την εμπορική εφαρμογή των καινοτομιών στην Ευρώπη εφόσον αναπτύσσονται για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες και επίγουσες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Και βέβαια, όπως και ο κ. Μπουζόη ανέφερε, έχω κατά νου και εγώ τα θέματα της υγείας και της βιώσιμης ανάπτυξης και συμφωνώ εδώ με τον εισηγητή που τονίζει αυτά τα θέματα στην έκθεσή του και ανέφερε και συγκεκριμένες ε, τροπολογίες ε, επί του θέματος. Όπως είπε και η κυρία Καπεσό, και αυτή είναι η ουσία του θέματος, είναι ο προϋπολογισμός ε, κάτι λιγότερο από 100, ε, ε, λιγότερο τέλος πάντων από ό,τι θα περιμέναμε. Είπατε, είπε ο εισηγητής 20 δισεκατομμύρια παραπάνω, αλλά η έκθεση Λαμή μιλούσε για 160 και εμείς εδώ μιλάμε για 120. Είμαστε μακριά από το στόχο του 3% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ, Άρα αυτό είναι κάτι που θα το τονίσουμε στις τροπολογίες μας. Τέλος, κάτι που θέλω να διευκρινίσουμε με τον εισηγητή, που είναι λίγο τεχνικό θέμα, αν σωστά σας παρακολούθησα, μιλάτε για τον τομέα παρέμβασης για τις τεχνολογίες της υγείας και μιλάτε για τον πόλο της υγείας και μια μετάβαση στον ψηφιακό πόλο. Μήπως με αυτή τη μετάβαση μπαίνουμε σε θέματα τεχνολογίας που είναι πολύ ευρύτερα και ίσως διαχέεται το ενδιαφέρον σε σχέση με τα καθαρά θέματα υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Κανείς άλλος που θέλει το λόγο? Αν όχι, θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή, τον κύριο Μακέιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, την οποία χαιρετίζουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Μπουζόη που έκανε μια χρήσιμη εργασία. Είχαμε και χρήσιμη συζήτηση και διευκρινίστηκαν ορισμένα θέματα. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι εν συντομία τρία-τέσσερα λεπτά να σας μιλήσω για το πώς αντιλαμβανόμαστε μερικές από τις τροπολογίες, μερικά γενικά σημεία και μερικά πιο ειδικά ειδικές αιτιολογικές σκέψεις ή άρθρα. Γενικό σημείο είναι όλες οι τροπολογίες που είναι γενικής φύσης, που μιλάνε για κατεξουσιοδότηση, πράξης, προϋπολογισμό, Ξέρουμε ότι είναι ε, ε, είναι το πακέτο το τελικό. Βεβαίως θέλουμε υψηλότερο προϋπολογισμό, αλλά στο τελικό στάδιο των συζητήσεων θα συζητηθεί το θέμα. Δεν θα ε, σχολιάσω το θέμα αυτό. Ίσως μερικές από τις τροπολογίες ε, οδηγούν σε τεχνική συζήτηση. Έχουμε μια τεχνική συνεδρία σήμερα το απόγευμα, οπότε θα διευκρινιστούν μερικά θέματα. Υπάρχουν κάποιες επαναλήψεις, μερικές τροπολογίες επαναλαμβάνουν ε, ορισμένες αντιλήψεις, ορισμένες ιδέες στην αηφορία. Βεβαίως χαιρετίζουμε την αηφορία, αλλά ίσως να μην επαναλαμβάνεται τόσο συχνά. Επίσης, ε, ορισμένες τροπολογίες έχουν υπερβολικές λεπτομέρειες. Ίσως ορισμένες μπορούν να αναφέρονται στην διαδικασία ε, προγραμματισμού στρατηγικής σε περαιτέρω φάση. Υπάρχουν πολύ καλές ιδέες ε, και που είναι στις τροπολογίες, αλλά πολλές φορές ξεπερνούν το όριο ε, που ε, μπορεί να έχει ένα τέτοιο πρόβλημα, πρόγραμμα. Ε, καταλαβαίνουμε την πρόθεση. σε ορισμένα άρθρα ίσως επεκτείνονται πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει. Μερικές κρίσεις αξίας θεωρούνται ως αρνητική συνειρμή, συσχετισμοί ε, σχετικά με ορισμένε ε, πολιτικές. Άρα τώρα θα μπω ε, σε μερικές περισσότερες λεπτομέρειες. Στις αιτιολογικές σκέψεις, όπως είπα, χαιρετίζουμε ε, την, ε, ε, την υποστήριξη στην αηφορία, υποστηρίζουμε πλήρως. Στο τέλος του έτους θα υπάρξει ένα έγγραφο από τον κύριο Τίμερμανς από την Κομισιό. Ανοιχτή πρόσβαση προτείνεται σε πολλές τροπολογίες να μην, εγώ εμείς προτείνουμε να μην περιορίζεται ο ορισμός της πρόσβασης και έχουμε μια σύσταση σχετικά με το θέμα αυτό, για να υπάρχει κάποια συνέπεια για τα άρθρα τώρα. Και πάλι χαιρετίζουμε το γεγονός ότι υπογραμμίζεται η ε, σημασία των κοινωνικών αναγκών, της ε, συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Αυτό είναι ε, βασικό συστατικό στοιχείο της οικοδόμησης της Ευρώπης, της έρευνας και καινοτομίας. Ε, άρθρο 7, τροπολογία τι αποστολές είναι αν θέλετε μια από τις καινοτομίες του προγράμματος Horizon Ευρώπη Βρισκόμαστε σε διερευνητικό στάδιο, υπάρχουν ε, ενδιαφέρουσες ιδέες. Ο κύριος Μπουζόη ανέφερε τέτοιες ιδέες. Θα πρέπει να δούμε τους τομείς, θέλουμε να θέσουμε προτεραιότητες. Αυτό θα έρθει αργότερα σε μια συζήτηση που θα περιλαμβάνει τους ενδιαφερόμενους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μυστικά με τα θέματα IPR υπάρχουν ε, πολλές τροπολογίες, 17, ε, 19, θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη ευελιξία από ό,τι στο πρόγραμμα Horizon 2020. Υπάρχει μια πρόδρος ε, επίσης ευελιξία για τον προσδιορισμό των, των θεμάτων που ενδιαφέρουν, τροπολογίες. Υπάρχουν μερικές ε, επαναληπτικές τροπολογίες. Ο λόγο ε, και πάλι έχουμε ευελιξία, αλλά θα πρέπει επίσης να έχουμε και μια ημερομηνία για να κλείσουν τα πράγματα εν ευθέτω χρόνο. 34 υπάρχουν ορισμένες αναφορές. Δεν ξέρουμε αν εδώ είναι αποτελεσματικό. Δεν ξέρω. Βεβαίως αν είναι η πρόθεση εδώ ένα σημαντικό σημείο που μας απασχολεί επίσης είναι η μεταφορά στο κλάστερ 3 ε, το θέμα αυτό ε, στην, για να μεταφέρετε το θέμα το σημαντικό ε, στο ψηφιακό πόλο. Βλέπουμε μια συμπληρωματικότητα με το κλάστερ 3, το κλάστερ 1 που είναι για την υγεία, διότι το κλάστερ 3 είναι για την ανάπτυξη των τεχνολογιών, των πλατφορμών για γενικούς σκοπούς, αλλά είναι ουσιαστικό να διατηρήσουμε σε κάθε τομέα, σε κάθε κλάστερ ορισμένα ε, στοιχεία, διότι δεν ακούσαμε για την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών πρέπει να ενσωματώσουμε, να μεγιστοποιήσουμε ε, τη χρήση τους και εδώ έχουμε όλες αυτά τα κέντρα, τα κέντρα καινοτομίας θα πρέπει ίσως να διατηρηθεί στο κλάστερ 1. Σχετικά με τις ε, εταιρικέ σχέσεις, τροπολογία 28, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι ε, σημαντικό να τονιστεί το θέμα αυτό ε, και να υπάρξουν επίσης και συνεισφορές σε χρήμα, διότι πάρα πολλές φορές δεν γίνεται αυτό και νομίζω ότι σε χρήμα είναι ε, σημαντικά, σημαντικό στρατηγικά. Σχετικά με το ειδικά προγράμματα, ε, ορισμένα τεχνικά υπάρχουμε, έχει υπεριδίκευση, το κτό ε, είναι λόγος για μερικά θαλάσσια θέματα με λεπτομέρειες Αυτά θα συζητηθούν στην τεχνική συνεδρίαση. Χαιρετίζουμε την τροπολογία 9, την αναφορά στην κυκλική οικονομία, είναι ένα θέμα ευρύ. Έχουμε για τους πολίτες την επένδυση που κάνουμε. Έχουμε διάφορες διατάξεις σχετικά με την εκμετάλλευση, τα αποτέλεσμα, σημείο 6 ίσως εδώ. Ίσως υπάρχει κάποια ένσταση με μερικά θέματα, τα τροπολογία 18 αναφέρονται ε, αναφέρεται η ασθένεια, ο καρκίνος. Ξέρουμε τη σημασία της ασθένειας αυτής για τον ε, την κοινωνία, αλλά ίσως τον αναφέρεται ειδικά αυτή η ασθένεια, ίσως να είναι αντιπαραγωγικό. Ίσως ε, να πούμε μη μεταδοτικές ασθένειες. Ε, το καρκίνος είναι τέτοια ασθένεια. Ίσως να έχουμε μια πιο γενική αναφορά. τροπολογία 23 Υπάρχει ρητή αναφορά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν είναι καλή νομοθετική πρακτική να περιλαμβάνονται άλλοι οργανισμοί με το όνομά τους, διότι δεν έχουμε ε, κανένα μοχλό ε, αν θέλετε, ίσως αυτό να αποφευχθεί. Και για να κλείσω, Τροπολογία 48. Θα πρέπει αυτή η αναφορά να γίνεται στο κλάστερ 4 διότι αυτή είναι σε κρίση, διότι αυτό αναφέρεται στην συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και ίσως να μπει σε άλλο πλαίσιο. Καλές ιδέες του εισηγητή και πάλι και τους ευρωβουλευτές και ίσως το πρόγραμμα αυτό θα είναι ακόμα καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much now. Ευχαριστούμε πολύ. Ξανά ο λόγος στον κύριο Μπουζόη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομος θα είμαι. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Καπεζόν, σας ευχαριστώ για τη θετική σας αντιμετώπιση και για την πρότασή σας, για τις προτάσεις που υποβάλλετε. Θα περιμένω τις τροπολογίες σας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ε, μικρό ποσοστό ε, των ε, προγραμμάτων ήταν επιλέξιμα και μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με το Horizon 2020, άρα είναι θετικό να κάνουμε το επόμενο βήμα για το επόμενο πρόγραμμα. Σχετικά με τις εθνικές προτεραιότητες και το Ηνωμένο Βασίλειο και το Brexit, είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε το αν θα παραμείνουν στο πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οι συμμετέχοντες ε, στη χρηματοδότηση και στην ε, δυνατότητα να έχουν χρήματα από αυτό το πρόγραμμα. Προς την κυρία Ρίσταλ να πω ότι συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο. Ο σύνθετος χαρακτήρας ε, και τα, η διοικητική φραγμή είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε και αναφέρατε τον προϋπολογισμό. Και γι' αυτό πρότεινα να μεταφέρουμε ε, ε, αυτά τα οποία αναφέρονται στον ψηφιακό τομέα να μεταφερθούν στον τομέα της υγείας. Αυτό θα αυξήσει τον προπολογισμό τη υγεία και πρότεινα δύο λύσει. Πρώτον, να αυξηθεί ο προπολογισμό για αυτό το κλάστερ, για αυτή τη θεματική ομάδα, αλλά πρέπει να αυξηθεί και ο προπολογισμό ε, του προγράμματο συνολικά και αυτό δεν θα είναι απόφαση που να πω στη δική μας Επιτροπή. Θα πρέπει να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πρόκειται για μια σημαντική αύξηση. Κάτι άλλο θα πρέπει να μειωθεί. Η άλλη λύση θα ήταν να αφήσουμε περισσότερο χώρο ε, για τις αποστολές για τα θέματα που είναι καθαρά θέματα υγείας και να μεταφέρουμε μόνο αυτά τα έργα υγείας που έχουν σχέση με ψηφιακές λύσεις. Αυτά να μεταφερθούν σε ένα άλλο κλάστερ, μια άλλη θεματική ομάδα, αφήνοντας χωριστά αυτά που είναι καθαρά θέματα υγείας. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα εδώ. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις τεχνικές πληροφορίες που μας έχουν δώσει. Σήμερα θα ακολουθήσει μια τεχνική συνάντηση και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με πολλές συναντήσεις. Σημείωσα κάποιες παρατηρήσεις σας και έχετε δίκιο, ίσως κάποιες τροπολογίες είναι υπερβολικά λεπτομερείς και το σημείο σχετικά με την ΠΟΗ δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να μπει σε ένα νομοθετικό κείμενο. Έχετε δίκιο. Για τον καρκίνο πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια, σημαντι... μια σημαντική μνήα, επιμένω, και να γίνει μια σχετική ε, αποστολή, καταλαβαίνοντας βέβαια ότι πρέπει να ε, δώσουμε λεπτομέρειες και να είμαστε και σε επαφή με όλους τους ενδιαφερόμενους. Σε ένα νομοθετικό κείμενο δεν μπορούμε να βάλουμε μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας και ίσως κάποιες προτεραιότητες μπορούν να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον βεβαίως συμφωνήσουν και τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό πιστεύω θα δώσει ένα πολιτικό μήνυμα σε σχέση με το πρόγραμμα Ορίζων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπουτσόη για την παρουσίαση και για την ε, έκθεση. 5 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Ε, στην συνεδρία 11 Οκτωβρίου στην Ένβη θα γίνει η ψηφοφορία. Και τώρα, το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Εξετάζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης και δίνω το λόγο στον εισηγητή κύριο Πιέκα. Ευχαριστώ πολύ. Το έγγραφο αυτό εξετάζει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά είναι δύσκολο ε, να αφήσουμε απ' έξω τον τεράστιο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Μιλάμε για ένα τομέα που αποτελεί επανάσταση και στην τεχνολογία και στην κοινωνική συμπεριφορά και μια ε, προφανώς δεοντολογική επανάσταση. Και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε τα κατάλληλα έγγραφα τεκμηρίωσης για να εξηγήσουμε προς ποια κατεύθυνση κινούμεθα στους τομείς ε, της υγειονομικής περίθαλψης, της τεχνολογίας της υγείας, ε, σε προγράμματα ε, που αφορούν ανακάλυψη φαρμάκων και ξέρουμε ότι η ρομποτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική, παραδείγματο χάρη, και ε, αναπτύσσουμε μια νέα προοπτική, λαμβάνοντας υπόψη και την ε, γύρανση της κοινωνίας μας. Ε, η υγεία είναι ένας τομέας που ε, στο μέλλον θα τύχει ιδιαίτερη ε, σημασία γιατί η ρομποτική θα μπορέσει να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με αναπηρίε. Ε, και μιλάμε για μια επανάσταση στον τομέα των τεχνολογιών υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχουν βέβαια ηθικοί προβληματισμοί σχετικά με την αυτονομία των ρομπότ και τον αντίκτυπό τους στη σχεση γιατρου ιατρού-ασθενή. Ε, θέλουμε να ξέρουμε ποιος ε, θα έχει την εποπτεία ε, των ρομπότ. Και για τους ασθενείς τους ίδιους αυτό θα αποτελέσει μια πρόκληση για το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τον τομέα αυτό, να φροντίσουμε το γενικότερο πλαίσιο και η δράση την οποία πρέπει εμείς να αναλάβουμε συνίσταται στα εξή. Θέλουμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να καταρτήσει ένα σχέδιο δράσης, όχι μόνο για τώρα, αλλά και για το μέλλον, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη έχουμε αυτοκίνητα τα οποία μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς οδηγούς ε, στους δρόμους των πόλεών μας και ήδη γίνονται δοκιμές ε, χωρίς ε, ανθρώπινη συμμετοχή. είναι διαδικασίες τις οποίες πρέπει συνεχώς να παρακολουθούμε. Η δυναμική της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής σίγουρα θα έχει επιπτώσεις και στα νομικά πλαίσια που πρέπει να ισχύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα υιοθετήσαμε μία έκθεση για ιατρικές συσκευές. Όταν χρησιμοποιούνται ρομπότ στην ιατρική ή όταν ε, ένα ρομπότ αντικαθιστά ε, ένα νοσηλευτή. Πρέπει να δούμε από νομικής πλευράς αν ε, είναι μια συσκευή, μια ιατρική συσκευή ή κάτι παραπάνω. Ακόμη και η πρόσφατη λοιπόν αυτή νομοθεσία για τις ιατρικές συσκευές δεν είμαι βέβαιος ότι είναι προσαρμοσμένη σε αυτά τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας από πλευράς τεχνικής, τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν τέτοιες πρωτοβουλίες για να έχουμε σωστή εποπτεία του τομέα αυτού. Θα πρέπει στην προσπάθεια αυτή να επιλέξουμε ε, και μηχανικούς ε, και βιομηχανικούς και εκπροσώπους ε, του κλάδου, όπως επίσης και τους πολίτες. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε και το γενικότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο ούτως ώστε να μην είναι χαοτικό το πλαίσιο για τον τομέα της ιατρικής και της υγείας. τα νομικά θέματα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, γιατί ξέρουμε ότι γίνονται αγωγές κατά των ιατρών για ιατρικά σφάλματα. Τι θα γίνεται σε περίπτωση σφάλματος ε, ενός ρομπότ, Ποιο θα είναι υπεύθυνο ε, για ε, τέτοιου είδου σφάλματα. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ετοιμάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Στην παράγραφο 2 υπάρχει ένα σφάλμα το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε γιατί ε, πρέπει να διευκρινιστεί το κείμενο. Θα είναι μια τροπολογία του εισηγητού αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. τώρα στους γεώδης ο κύριος Μικολάσικ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Πιέκα για την πολύ καλή γνωμοδότηση για το θέμα αυτό που έχει εκθετικά αυξανόμενη σημασία. Σίγουρα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό με διεξοδικό και συγκεκριμένο τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ολοένα και αυξανόμενη παρουσία των νέων τεχνολογιών που βασίζονται στην τεχνική νοημοσύνη στη ζωή μας. Είναι ευθύνη μας ε, να παράσχουμε ε, σωστή διακυβέρνηση που θα βασίζεται σε ένα υγιές ε, νομοθετικό πλαίσιο σε συνεργασία με όλους τους αρμοδίους ενδιαφερομένους και πολίτες. Θυμάμαι μία επίσκεψη που κάναμε μελέτης ε, σε ένα ε, νοσοκομείο στη βέλγικη πόλη του Άλστ ε, πριν από κάποια χρόνια που μαζί με κάποιους συναδέλφους θαυμάσαμε ε, μία λαμπρή τεχνολογική ε, τελειότητα ενός ρομπότ Νταβίντσι στη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης. Ο χειρουργός χειριζόταν το μηχάνημα και μπόρεσε να κάνει μία επέμβαση με ιδιαίτερη ακρίβεια, κυρίως σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτό αφορά συγκεκριμένο αριθμό βέβαια χειρουργικών επεμβάσεων και όχι όλες τις επεμβάσεις. Η τεχνολογική πρόοδος ε, και τα ωφέλη ήταν αδιαμφισβήτητα. Όπω αναφέρεται και στη γνωμοδότηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική έχουν τεράστιες δυνατότητες, ε, ιδίω ε, στον τομέα της υγείας, που είναι ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά για όλους μας ε, και έχει εξίσου σημαντική σχέση με το περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων. Επομένως, ε, γνώσης ε, βάσει περίπλοκων δεδομένων και αναλύσεων των δεδομένων και εμπειρογνωμοσύνης ε, σίγουρα μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των διατάξεων της ασφάλειας των τροφίμων. Υποστηρίζω ακράδαντα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε τον Απρίλιο που τόνισε και την ευρωπαϊκή προσέγγιση για την όθηση στις επενδύσεις η οποία συνάδει και με τις ε, ηθικές δεντολογικές κατευθυντήριες γραμμές. Υποστηρίζω τη Συμμαχία της Τεχνητής Νοημοσύνης της Ευρώπης που θα καθορίσει και ε, κατευθυντήριες γραμμές περιδιοντολογίας ε, που θα βασίζεται και στη Χάρτα των Θεμολογικών Δικαιωμάτων και ε, θα συνεχίσει και την ε, Ευρωπαϊκή, όσα έκανε η Ευρωπαϊκή Ομάδα Ηθικής ε, στα τομέα της βιοτεχνολογίας και της επιστήμης. Η πρόσφατη δήλωση της ομάδας αυτής για την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τα αυτόνομα συστήματα είναι είπαν κατεπήγον να εξετάσουμε τα θέματα της ηθικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη, τη λεγόμενη αυτόνομη τεχνολογία, η οποία θα μπορούσε πιθανόν να δράσει χωρίς άμεσο έλεγχο ε, ανθρώπινου παράγοντα, ε, προς όφελος των ανθρώπων, αλλά και εις βάρος των ανθρώπων. Και βάσει αυτής της δήλωσης ε, θα ήθελα και εγώ να ζητήσω από την Επιτροπή μας να βασιστεί σε ηθικά στοιχεία που βασίζονται στην ανθρώπινη πρέπεια, στην ισότητα, στην αλληλεγγύη, στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη λογοδοσία, την ασφάλεια, την προστασία, την ε, ακαιρεότητα, τη σωματική και την ψυχική ε, και φυσικά την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όσον αφορά τα αυτόνομα ρομπότ. Ε, κάποιες συζητήσεις, ακόμα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρονται στην ιδέα ενός ειδικού νομικού καθεστώτος για τα ρομπότ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι διευκρινίζουμε ότι τα ρομπότ ανέκαθεν ήταν και θα συνεχίσουν να είναι απλώς αντικείμενα. Επομένως, ε, η ευθύνη είναι στα χέρια ε, του ανθρώπινου παράγοντα, είτε του κατασκευαστή είτε του χρήστη και δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα ε, του δίθεν ανθρωπισμού ε, με στόχο απλώς να αποδεσμεύσουμε τους ανθρώπους από την τεχνολογική πρόοδο. Είμαι βέβαιος ότι μαζί θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες ε, δεντεολογικές και νομικές ε, στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική και να βρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη γραμμή. Προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία για το θέμα αυτό και περιμένω να έχουμε καλές και επικοδομητικέ τροπολογίες για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζεντήλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Δεν θα ξαναπώ τα όσα ακούσαμε ήδη και την αξιολόγηση της ποιότητας του κειμένου με το οποίο συμφωνώ, αλλά Θα ήθελα όλοι μας να καταλάβουμε και πόσο σημαντική είναι η συζήτηση που γίνεται μέσω αυτής της γνωμοδότησης στην Επιτροπή αλλά και στην αξιολόγηση των κρατών μελών και της διεθνούς γνώμης. Η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες ε, σήμερα μπορούν ε, να συνοδεύσουν μια διαδικασία ποιοτική ε, και να δώσουν μια απάντηση στη, ε, στο αίτημα της υγείας ε, και πώς μπορούμε μέσω αυτού να ανοίξουμε νέους χώρους για την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα των ε, εθνικών συστημάτων υγείας. Δεν θα σας πω εδώ στοιχεία και αξιολογήσεις, δεν χρειάζεται. Ξεκινάει μια διαδικασία στην οποία τα αριθμητικά στοιχεία θα αυξηθούν εκθετικά και όλα αυτά θα συνοδεύονται από το αίτημα της υγείας, το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε χωρίς την τεχνολογική καινοτομία. Είναι πολύ σημαντικό το κόστος για την υγεία. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί, για παράδειγμα, οι οποίοι δεν μπορούν να αυτοσυντηρηθούν ε, και πάσχουν από χρόνιες ασθένειες ε, και ζητούν να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο είναι κοινό για τα κράτη-μέλη. Η καινοτομία λοιπόν, αλλά με μεγάλη ευφυΐα είναι αυτή που θα βοηθήσει. Δηλαδή το να φεθούμε απλώς στην τεχνολογία χωρίς ε, να διατηρήσουμε και να προφυλάξουμε και το ανθρώπινο και ατομικό προφίλ κάποιου μπορεί τελικά να περιορίσει ε, μια εξαιρετική ευκαιρία. Μαζί λοιπόν με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, αλλά και με τη στήριξη των επιχειρήσεων βεβαίως, που προφανώς ε, έχουν χίλιους λόγους να πειραματίζονται στον τομέα αυτό, να μην ξεχνάμε δε ότι στο συγκεκριμένο τομέα μπορούμε να προσφέρουμε και ε, ευκαιρίες εργασίες ε, για κατάλληλες δεξιότητες οι οποίες είναι επιθεματές στον τομέα της υγείας, στον τομέα της συλλογής των δεδομένων, βάσει των οποίων θα ε, καθορίσουμε από εκεί και πέρα διαδικασίες πρόληψης, θεραπείας ε, ε, και συγκεκριμένη φροντίδα που θα βασίζεται ε, σε ε, συγκεκριμένα αιτήματα. Παραδείγματο χάρη, εμβολιασμό. Πώ μπορεί η συλλαγή των δεδομένων να μα βοηθήσει να προσανατολίσουμε τι πολιτικέ επιλογέ στον τομέα ε, των εμβολίων, για παράδειγμα για ηλικιωμένου ή για άτομα τα οποία ζουν σε δυσάρεστες καταστάσεις ακόμα και σε γεωγραφική έκταση, ανθρώπους δηλαδή που ζουν σε πολύ απομονωμένες περιοχές και πώς μπορούμε να πούμε, και πάντα αυτό σε αναφορά το κόστος, θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση των δαπανών. Για παράδειγμα, της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, στην πρόληψη της έλλειψης προσανατολισμού σε κάποιες ε, χρόνιες παθήσεις και πώς αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιορίσει τις δημόσιες διαπάνες, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, εάν ε, ε, ε υπάρχει κατάλληλη χρήση φαρμάκων και πώς μέσω της ε, ε τεχνολογίας, για παράδειγμα, ε, μια κάψουλα που όταν δεν ε, τη λάβει κάποιος ε, στέλνει μήνυμα ότι κάποιο ξέχασε να πάρει το χάπι του. Πώς μπορούμε έτσι να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων και να ζουν όλοι πάνω από, 100, πάνω από 65 πριν από το θάνατό τους. Ο κύριο Πέκ. Ο κύριο Έκ, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είναι αδιαμφισβητητό ότι στο μέλλον η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει το μέλλον σε πάρα πολλούς τομείς. Στην ιατρική, στην έρευνα, στην οδική κυκλοφορία, ακόμη και στον τομέα των κατασκευών. Εδώ έχουμε θέματα δεοντολογίας και θα είναι πολύ θετικό όταν ε, με υπευθυνότητα αντιμετωπίσουμε τις νέες αυτές τεχνολογίες. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική σίγουρα θα προκαλέσουν και κάποιες παράπλευρες ζημίες. Οι αρνητικές επιπτώσεις που δυστυχώς είναι αναπόφευκτες θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν μέσω μιας υπεύθυνης πολιτικής. Ο πολιτικός έλεγχος λοιπόν και η πολιτική εποπτεία θα είναι απαραίτητη. Θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση και να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική ε, μόνο εφόσον αναλάβουμε τις ευθύνες μας και δεν επιτρέψουμε να ε, εξαπλωθούν ε, εσφαλμένες ειδήσει και εσφαλμένε ε, ε, ε, απόψεις σε πολλές περιοχές του κόσμου. Κατά τη γνώμη μου, ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε τις παράπλευρες ζημίες είναι μια αυστηρή πολιτική εποπτείας διότι επιμένουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει μια σημαντική πρόοδο, την οποία πρέπει να προστατεύσουμε. Χαίρομαι για τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν να συζητήσουμε με τους αγαπητούς συναδέλφους αυτό το καυτό θέμα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζολίνιο. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντίθετα με τα όσα είπε ο συνάδελφος, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο κλειδί της συζήτησης σε αυτό το κοινοβούλιο, διότι εμείς αντιπροσωπεύουμε την ευρωπαϊκή κοινωνία και αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί στην εξέλιξη των κοινωνιών μας και αυτές οι αλλαγές τεχνολογικές θα πρέπει να εξυπηρετούν τα άτομα ε, κυρίως στον τομέα της υγείας, αλλά αυτό ισχύει σε όλους ε, τους τομείς της κοινωνικής ε, ζωής για να μπορέσουμε να ευνοήσουμε με μεγαλύτερη σύγκληση ευρωπαϊκή για να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες στα άτομα στις περιφέρειες και γενικά θα πρέπει να έχουμε ένα μοντέλο ψηφιακής οικονομίας χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών μας αξιών των κοινών μας αξιών και των προτεραιοτήτων μας. Υπάρχουν τεχνολογικές διαστάσεις, οικονομικές, ηθικές. Αυτά λέχθηκαν. Αλλά αν ζήτησα τον λόγο είναι επειδή είμαι σκιώδης εισηγητής για το πρόγραμμα ψηφιακής Ευρώπης και ήθελα να διευκρινίσω ότι το πρόγραμμα αυτό με 2 δισεκατομμύρια ε, ε, ευρώ σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, για τους πολίτες και θα πρέπει να εργαστούμε με τρόπο πάρα πολύ αποτελεσματικό. Θα εντάξουμε την ε, πρωτοβουλία αυτή στο πρόγραμμα ψηφιακής Ευρώπης με συγκεκριμένα προγράμματα, με το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη για να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από τις αλλαγές αυτές για να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε να αντιμετωπίσαμε. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. επικεφαλής της Μονάδας Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομπητικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή για αυτήν το σχέδιο γνωμοδότησης, διότι θέτει ορισμένα σημαντικά σημεία και θέματα που εμείς στην Κομισιόν σκεπτόμαστε ότι είναι χρήσιμα και τα οποία λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά πάρα πολλά σημεία που αναφέρονται στο κείμενο αυτό ε, έχουν συνάδουν με τη σκέψη της Κομισιό, έτσι όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση ε, για την τεχνητή ε, νοημοσύνη που υιοθετήθηκε στις 25 Απριλίου αυτού του έτους. Και δίνοντας ένα παράδειγμα θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό βεβαίως να έχουμε αυξημένη χρηματοδότηση όπως είπε προηγούμενος ομιλητής, διότι πώς αυτή η τεχνολογία στο μέλλον θα έχει σημαντική επίπτωση στη ζωή μας, στην εργασία μας και σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για τα νομικά θέματα, τα ηθικά θέματα, τα θέματα υπευθυνότητας, ε, το θέμα της ανάπτυξης, της ε, τεχνολογίας και Όντως, το κλειδί ε, στην προσέγγιση της Κομισιό, έτσι όπως το παρουσιάσαμε, είναι μια προσέγγιση ολιστική για να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση που να διακρίνεται από αυτό που παρουσιάζεται στην Ασία και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Και εδώ είναι σημαντικό να διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης, δηλαδή ότι λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά και τις μη ε, τεχνολογικές ε, πτυχές. Η πρωτόβουλη αυτή δεν έχει μόνο συστατικά τεχνολογικά, αλλά και άλλα που δεν είναι τεχνολογικά. Έχουμε λοιπόν να δούμε πώς θα ετοιμαστούμε για τα κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που θα προκαλέσει αυτή, ε, αυτή η τεχνολογία. Θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ε, ισχυρό ε, στην Ευρώπη μέσα στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 ε, και ε, για την επόμενο πρόγραμμα ψηφιακής Ευρώπης και το πρόγραμμα Ορίζων Ευρώπης στα πλαίσια του επομένου ε, πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε ειδικά μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία συζητούνται επίσης. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με συστήματα δοκιμής νέων τεχνολογιών, είναι λεπτομέρειες που θα πρέπει να μας επιτρέψουν να έχουμε ένα οικοσύστημα ε, ευρωπαϊκό τεχνητής νοημοσύνης που να είναι δυνατό. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να παρακολουθούμε τις εξελίξεις αυτής της τεχνολογίας και να λάβουμε υπόψη για να δούμε εάν η εφιστάμενη νομοθεσία και αυτό αναφέρθηκε υπάρχει ήδη εφιστάμενη νομοθεσία για αυτήν την τεχνολογία να δούμε αν είναι κατάλληλη για το στόχο μας και αν πρέπει να αναθεωρηθεί ε, θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε την εξέλιξη ε, από κοντά και να δούμε αν χρειάζονται αλλαγές νομοθετικές. Ε, θέλουμε αποτελεσματικά να έχουμε μια προσέγγιση που να ωφελεί τα, τους πολίτες και την κοινωνία στο σύνολό της, στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν μέτρα, κυρίως όσον αφορά την, τα ηθικά και ε, νομικά θέματα και Θέλουμε δύο αποτελέσματα, να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές ως προς την, τα ηθικά σημεία και δεύτερον ε, να έχουμε ε, συστάσεις. Το πρώτο σχέδιο θα πρέπει να υπάρχει στο τέλος του έτους και μια πιο πλήρη εκδοχή το επόμενο έτος αυτό το, η ομάδα υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων ε, περιλαμβάνει πανεπιστημιακούς, ε, την βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών, διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων που αντιπροσωπεύονται σε αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Και αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων αλληλεπιδρά ε, με την AI Alliance που είναι ένα φόρουμ ε, πολλαπλό, πολλαπλών ενδιαφερομένων που ασχολείται, υπάρχουν εκατοντάδες μέλη, διάφορες απόψεις εκφράζονται, όλοι μπορούν να, ε, να συμμετάσχουν σε αυτήν την ε, συμμαχία, σε αυτό το φόρουμ και τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα υποβληθούν στην ομάδα υψηλού επίπεδου. Επίσης για τα θέματα υποφθηνότητας έχουμε μια ομάδα, ένα από τα μέτρα στην ανακοίνωση είναι ότι θα υπάρχει μια έκθεση πιο ε, περιεκτική για τα θέματα υποφθηνότητας και συμπεράσματα σε σχέση με αυτήν την τεχνολογία. Θα έχουμε την ανακοίνωση το επόμενο έτος. Αυτά είναι μερικά από τα μέτρα τα πιο συγκεκριμένα τα οποία θα μας επιτρέψουν να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη και τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν εδώ σε αυτή την αίθουσα αντανακλούν την σημασία που ε, έχει αυτό το θέμα και που έχει και για την Κομισιό αυτή η ανακοίνηση. Υπάρχει ζήτηση μεγάλη για μια καλή προσέγγιση, ανθρώπινη προσέγγιση για το θέμα τεχνητής νοημοσύνης όχι μόνο από τους πολίτες αλλά και από τις επιχειρήσεις για μια τέτοια προσέγγιση που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανθρώπινες πτυχές, τις συνέπειες της τεχνολογίας, διότι πρέπει να παράγεται αυτή η τεχνολογία μέσα σε ένα περιβάλλον που θα είναι προς όφελος όλων και θα επιτρέπει ε, στους Ευρωπαίους να επωφεληθούν μακροπρόθεσμα το μέγιστο από αυτήν την τεχνολογία. Θα ήθελα να τονίσω κάτι κλείνοντας σχετικά με την γνωμοδότηση. Τα κράτη-μέλη έχουν, ε, συντάσσουμε με τα κράτη-μέλη ένα συντονισμένο σχέδιο μέχρι το τέλος του έτους και υπήρξε μια δήλωση που από 24 μέλη και την τεχνολογία έχει υπογραφεί. Αυτή η τεχνολογία έχει οθετηθεί από όλα τα κράτη-μέλη τώρα και την Ορβηγία βεβαίως. Έχουμε λοιπόν μια βάση, τη βάση των κρατών μελών για αυτήν την τεχνολογία. Ε, ένα πράγμα που ανέφερα και είναι προφανές το θέμα της εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας προσέγγιση που θα λάβει υπόψη όλα αυτά τα τεχνικά, νομικά και ηθικά άτομα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Κατανοώ ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι σύντομη, αυτή είναι η διαδικασία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, έλαβε υπόψη το θέμα αυτό και έλαβε υπόψη τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ε, ξέρουμε ότι έχει κατακτήσει όλους τους τομείς της ζωής μας, αλλά ε, στην ιατρική, στην υγεία, ε, είναι, έχει σχέση με την ιδιωτικότητα. Γι' αυτό και η ασφάλεια είναι ε, σημαντική για το μέλλον. Ως πολίτης, ως ευρωβουλευτής, ε, ανησυχώ, είμαι επιφυλακτικός διότι έχω ανατραφεί σε ένα κλίμα όπου όλα ήταν προσανατολισμένα προς τον άνθρωπο αλλά όλα αλλάζουν τώρα και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει έλλειψη ανθρωπισμού στους πληθυσμούς μας και στις, στην υγειονομική φροντίδα. Ελπίζω ότι έχω δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ όλους για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση τροπολογίας 5 ε, Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε τον Νοέμβριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη συνεδρίαση στο Στρασβούργο.